Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε. Γιατί όπως γνωρίζετε έχουμε μια πολύ σημαντική ακρόαση με θέμα το Brexit και καλό θα ήταν να έχουμε αρκετό χρόνο για να τις αφιερώσουμε. Γι' αυτό και θεωρώ ότι καλό θα ήταν σιγά σιγά να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας κάποια εισαγωγικά πρώτα να έχουν το χρόνο να έρθουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Ε, ως προς την ημερήσια διάταξη υπάρχουν παρατηρήσεις, όχι από ό,τι βλέπω, οπότε την εγκρίνουμε. Καταρχήν ε, να σας υπενθυμίσω ότι αναμεταδίδεται στο διαδίκτυο η συνεδρίασή μας και έχουμε διερμηνία σε 16 γλώσσες. 15 πια, γιατί δεν υπάρχουν τα δανέζικα. Τώρα, αν δεν υποβληθούν παρατηρήσεις για τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Δευτέρα Οκτωβρίου και 9 η και 10 η Οκτωβρίου μέχρι το τέλος συνεδρία θα θεωρηθούν ως συγκεκριμένα τα σχετικά πρακτικά. Περνάμε στο σημείο 4. Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Θα ψηφίσουμε τη σχετική γνωμοδότηση. Έχουμε 66 τροπολογίες για το θέμα αυτό. Στόχο έχει πρωτοβουλία την ε, μίση των νέων ε, στον εθελοντισμό και την εξασφάλιση δυνατότητας ε, να απασχολούνται σε έργα που ωφελούν τις κοινότητες και τις φλώσεις της Ευρώπης. Αρμόδια καθήλου επιτροπή είναι η Επιτροπή Πολιτισμού και Περιβάλλοντος. Στα πλαίσια της διαδικασίας εφαρμόστηκε το άρθρο 53 παράγραφος 4 προκειμένου να αναλάβουμε τη γνωμοδότηση. Πρόκειται για μια καινούργια διαδικασία και ουσιαστικά δεν έχουμε πραγματικό συντάκτη γνωμοδότησης, ούτε σχέδιο γνωμοδότησης κανονικό. Έχουν όμως κατατεθεί τροπολογίες και την γνωμοδότηση την υποβάλλει ο πρόεδρος ε, της Επιτροπής εν είδη συντάκτης γνωμοδότησης. Αυτά ως προς τα διαδικαστικά. Όπως σας είπα, αρμόδια κατ' επιτροπή είναι η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Και δεν ξέρουμε πότε θα ψηφιστεί η έκθεση αυτή στην Ολομέλεια. Αλλά ας περάσουμε στην ψηφοφορία μας. γιατί δεν βλέπω ερωτήσεις, απορίες από την αίθουσα. Τροπολογία 34. 34 παρακαλώ ποιος είναι υπέρ. Διανατάσσω στις χειρός. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 33. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 31 υπέρ. Εγκρίνεται. 32 υπέρ. Εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά, απορρίπτεται. 36 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 37 υπέρ, εγκρίνεται. 38 υπέρ, εγκρίνεται. 39 υπέρ, εγκρίνεται. 40 υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος, παρακαλώ για να το άρχεται η ψηφοφορία για να ελέγξουμε το αποτέλεσμα τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά μόνο τροπολογία 41 ποιος είναι υπέρ κατά απορρίπτεται 42 υπέρ εγκρίνεται 43 υπέρ εγκρίνεται 44 υπέρ κατά ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχιτη ψηφοφορία παρακαλώ τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται συγχαρητήρια στον εισηγητή που απουσιάζει όμως τροπολογία 45 ποιος είναι υπέρ εγκρίνεται 46 υπέρ εγκρίνεται 47 υπέρ εγκρίνεται. 48 υπέρ, εγκρίνεται. 49 υπέρ, εγκρίνεται. 50 υπέρ, εγκρίνεται. 51 υπέρ, εγκρίνεται. 52 υπέρ, εγκρίνεται. 53 υπέρ, κατά Ηλεκτρονικό έλεγχο για την τροπολογία 53. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 54 υπέρ. Εγκρίνεται. 55 υπέρ. Εγκρίνεται. 56 υπέρ. Εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος και για την 57 άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 58 υπέρ. Εγκρίνεται. 59 υπέρ. Εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 64 υπέρ, εγκρίνεται. 65 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 66 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ, εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ, εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ, εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ εγκρίνεται. 6 υπέρ εγκρίνεται. 7 υπέρ εγκρίνεται. 8 υπέρ εγκρίνεται. 9 υπέρ εγκρίνεται. 10 υπέρ εγκρίνεται. 11 υπέρ εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ εγκρίνεται. 13 υπέρ ε, κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14 υπέρ κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Μάλλον απορρίπτεται. Τέλος ψηφοφορίας. Όντως. Απορρίπτεται. Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 16. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 17 υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 23 και 24 υπέρ εγκρίνεται. 25 υπέρ, εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τις τροπολογίες 23 και 24, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνονται. Τροπολογία 25 υπέρ 25 εγκρίνεται. 26 υπέρ. Εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 28 υπέρ. Καταπίπτει 28. Πάμε στην 30 κατευθείαν. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Οπότε ψηφίζουμε το σύνολο της γνωμοδότησης όπως έχει τροποποιηθεί. Άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ποιο να ευχαριστήσω. Άντε τους ε, συντάκτες των τροπολογιών, γιατί ε, συντάκτη γνωμοδότησης δεν είχαμε. Σας ευχαριστώ πάντως για την άρτια διεξαγωγή της ψηφοφορίας και περνάμε στο σημείο 5. Έχουμε το ζήτημα για το οποίο αρμόδιος είναι ο κύριος Ιβάν Γιάκοφτσίτς, τον οποίο και καλωσορίζω θερμότατα. Χαίρομαι που θα υποβάλουμε σχετική γνωμοδότηση. Καταρχήν να θυμηθούμε το εξαιρετικό ελαιόλαδο της Ίστριας. Άρα να δώσω κατευθείαν το λόγο στον εισηγητή μας, που είναι και ο πλέον αρμόδιος για να μας κάνει την ενημέρωση για το θέμα αυτό. Κύριε Γιακόφτσιτς, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου, στο μέτρο που ακούγεται ε, θόρυβος ακόμη στην αίθουσα, να ευχαριστήσω και εσάς και τα μέλη της Επιτροπής για την εμπιστοσύνη που δείξαν αναθέτοντάς μου αυτή την γνωμοδότηση για τη σύνοψη, σύναψη Διεθνούς Συμφωνίας ε, για του 2015 για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζεις ελιές. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου είναι η αρμόδια καθήλη επιτροπή για το θέμα αυτό. Η Επιτροπή Ίντα δηλαδή θα συντάξει ε, την έκθεση με τη γνώμη για τη σύναψη αυτής της ε, συμφωνίας και μάλιστα η Επιτροπή Ίντα θα αποφασίσει μετά από μας. Αυτό που είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε είναι ότι η όλη διαδικασία κόλλησε στις σχέσεις Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και κυρίως ε, ε, στο άρθρο που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το άρθρο 4, για τη διαδικασία στην σύναψη αυτής της Διεθνούς Συμφωνίας ελπίζω αυτό που δεν συνέβη μέχρι στιγμής να γίνει, δηλαδή να διαθετήσουν τις διαφορές τους και τα διλήμματά τους ε, το Συμβούλιο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η γνωμοδότησή μας ουσιαστικά δίνει τη θετική μας γνώμη, την ε, συνένεσή μας ε, για το θέμα αυτό και καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να συνάψουν αυτή τη Διεθνή Συμφωνία για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές. Αυτή είναι η ουσία της γνωμοδότης ουσιαστικά. Ε, μπορούμε να συντάξουμε τροπολογίες και να είμαστε και κατά. Μόνο αυτό μπορούμε να κάνουμε ουσιαστικά από νομική άποψη. Μια όμως και κάθε γνωμοδότηση έχει και την εισαγωγή της και ένα είδος σύντομης αιτιολόγησης, θα ήθελα και στη δική μου γνωμοδότηση να σας υπενθυμίσω αυτά που έχουν συμβεί μέχρι στιγμής, από το 2013 δηλαδή, μέχρι το 2017 ουσιαστικά, μέχρι τη σήμερα ημέρα δηλαδή. Και να σας... Ε, ε, υποβάλλω τι προτάσει μου που προκάλεσε μια πολύ θετική κατά τη γνώμη μου συζήτηση. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή τη στιγμή, τη στιγμή δηλαδή που συζητάμε και πάλι για τη διεθνή αυτή συμφωνία που έχει μια καινοτομία σχέση με τις προηγούμενες διεθνείς συμφωνίες. Και εγώ προτείνω σε αυτή την σύντομη μου αιτιολόγηση να προσπαθήσουμε να ρυθμίσουμε καλύτερα την αγορά ελαιολάδου από ό,τι σήμερα. Και γι' αυτό για την προστασία δηλαδή των παραγωγών και κυρίως για την προστασία των καταναλωτών, προτείνω η Επιτροπή να λάβει υπόψη την κατάσταση στην αγορά ελαιολάδου και να βρούμε τρόπο να θεσπίσουμε μια νέα κατηγορία για το ελαιόλαδο. Την ε, κατηγορία αρίστης ποιότητας, δηλαδή αυτό που εγώ αποκαλώ premium εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και πολλή παραγωγή από τη Μεσόγειο, παραγωγή ελαιολάδου, κυρίως από μεσογειακές χώρες που είναι ε, χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παράγουν τέτοιο πρέμιο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο που υπολογίζουμε ότι είναι περίπου το 15% της παγκόσμιας παραγωγής, αυτό που δηλαδή που πραγματικά αξίζει τον προσδιορισμό του πρέμιου εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου. Σε αυτή ε, μέχρι στιγμή αυτή την κατηγορία δεν την έχουμε. Έχουμε το, την ανώτερη κατηγορία του εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Όμω είναι τόσο ε, ποικιλόμορφη αυτή η κατηγορία και τόσο ευρύ το φάσμα των τιμών, τι να σας πω, μπορείτε με 4 ευρώ να βρείτε σήμερα στην αγορά εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο μέχρι 30 ευρώ. Είναι τεράστια η ψαλίδα των τιμών και η ποιότητα είναι ποικίλη. Νομίζω ότι έχει νόημα να θεσπίσουμε και μία νέα κατηγορία του πρέμιου εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, τιμώντα ε, τους παραγωγούς τέτοιου είδους ε, άριστου ελαιολάδου για να βοηθήσουμε και του καταναλωτές ε, να αντιληφθούν τις διαφορές στην ποιότητα. Νομίζω ότι είναι αξιέπαινη αυτή η πρωτοβουλία και μπορούμε να συζητήσουμε από αυτό. Εν κατακλείδη, θα ήθελα να πω ότι σήμερα πρέπει να αποφασίσουμε αν είμαστε υπέρ της σύναψης της Διεθνούς Συμφωνίας σχετικά με το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές του 2017. Εγώ είμαι υπέρ της σύναψης αυτής της συμφωνίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Γιακόφτσιτς. Ζήτησαν το λόγο κάποιοι συνάδελφοι. Κυρία Ράνς Γκαρσία πρώτα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς ο κύριος Βαλκάρσελ που είναι ο σκιώδης ηγητής ε, του ΕΛΚ για τη γνωμοδότηση αυτή χρειάστηκε να πάει στην Πράγα σε μια ε, συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και τον αντικαθιστώ εγώ. Ε, μάλιστα με τιμά ιδιαίτερα αυτό το θέμα γιατί και το ελαιόλαδο και οι επιτραπέζιες ελιές είναι για την Ισπανία ζήτημα κέρια σημασία. Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τις προσπάθειές του και ε, να μιλήσουμε για αυτή τη συμφωνία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί απλώς να γνωμοδοτήσει δίνοντας τη συνένεσή του ή όχι. Ουσιαστικά είναι τυπικό το θέμα του, της γνώμης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, ο εισηγητής στην αιτιολόγηση πρότεινε την θέσπιση μιας νέας κατηγορίας για το ελαιόλαδο που είναι το premium ε, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Και μας εξήγησε ο συντάκτης ότι αυτό είναι αίτημα των ίδιων των παραγωγών της Κροατίας. Η δική μας όμως παραγωγή από την Ισπανία το αντίθετο μας ζητούν. Μας λένε ότι ήδη αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα ε, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές και δεν μπορούν να κάνουν τη διαφοροποίηση μεταξύ του έξτρα παρθένου, του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου και του παρθένου ελαιολάδου. Τώρα αν προσθέσουμε και μία νέα κατηγορία με το premium εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο θα τους περδέψουμε ακόμη περισσότερο τους καταναλωτές μας. Αυτό ισχυρίζονται οι Ισπανοί παραγωγοί. Κατά τη γνώμη μας ε, δεν μας πείθουν τα επιχειρήματα ε, του κυρίου Γιακόφτσης, γιατί όπως ξέρετε στη Ισπανία έχουμε πολλά και πολύ ποιοτικά ε, ελαιόλαδα και μάλιστα μεγάλη παραγωγή. Και μάλιστα είχαμε και συνάδελφο ε, την κυρία Κλάρα Αγγελέα που ήταν σύμβουλος στην Ανταλουσία που είναι η μεγαλύτερη παραγωγός περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε θα ήθελα περισσότερες εξηγήσεις γιατί νομίζω ότι η πρόταση για τη θέσπιση μιας επιπλέον κατηγορίας για το ελαιόλαδο θα φέρει τα αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα που είναι η βοήθεια στους καταναλωτές να κάνουν τη διαφοροποίηση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντες. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ήθελα να ακούσω πρώτα τη συνάδελφο Αλιγκέρα, γιατί δεν έχουμε πολλέ έλειες στη Γερμανία. Επομένω, την ακολουθώ. Λέω και εγώ, στη Βαβαρία δεν είδα και πολλά ελαιόδεντρα, οι ε, Όπω Όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Ράς Γκαρσία. Ε, θα ήθελα να πω στον ε, εισηγητή μας ότι για την συμφωνία για το ελαιόλαδο δεν έχουμε πρόβλημα. Πολύ ευχαρίστω να συνενέσουμε, αλλά το να θεσπίσουμε μια νέα κατηγορία, ένα νέο προσδιορισμό για το ελαιόλαδο, αυτό είναι παρακινδυνευμένο. Γιατί ε, μας είπατε ότι το ζητούν οι ίδιοι οι παραγωγοί. Δεν ξέρω ποιοι παραγωγοί, γιατί τουλάχιστον στην πατρίδα μου, την Ισπανία, και τουλάχιστον στην περιφέρεια που εγώ γνωρίζω καλύτερα την Ανταλουσία, δεν είναι αυτό το αίτημα των παραγωγών. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μεγάλη σύγχυση για το καταναλωτή με την ύπαρξη πολλών ε, κατηγοριών ελαιολάδου. Και τα μεγάλα σούπερ μάρκετ ε, επηρεάζουν ε, ιδιαίτερα όχι μόνο την αλυσίδα παραγωγής αλλά και τον προσδιορισμό των τιμών. Και μάλιστα οι μεγάλες αλυσίδες διανομής χρησιμοποιούν και τις δικές τους κατηγορίες. Ήπιο, πικρό ελαιόλαδο, έντονο ουσιαστικά για να μπερδέψουν τον καταναλωτή και να μην ξέρει τι βρίσκεται πίσω από αυτό το ελαιόλαδο. Και υπάρχει ήδη σύγχυση στην αγορά. Και ο κλάδος, που γνωρίζω πολύ καλά, ισχυρίζεται ότι οι κατηγορίες είναι πολύ καλά προσδιορισμένες. Το να προσθέσουμε ακόμη μια νέα κατηγορία στο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ε, που είναι το καλύτερη ποιότητα ελαιόλαδο, μόνο σύγχυση θα μπορούσε να αυξήσει και να δημιουργήσει παρά να διευκρινίσει τα πράγματα. Σίγουρα υπάρχουν εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα με πολλέ και διάφορε τιμέ. Από 4 ευρώ το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο μέχρι 30 ευρώ. Αυτό όμω δεν έχει σχέση με τον κλάδο, δεν έχει σχέση με του παραγωγού, δεν έχει σχέση με του καλλιεργητέ. Ούτε υποφελούνται οι παραγωγή από αυτές τις διαφορές. Αυτό είναι θέμα των σούπερ μάρκετ και των διατροφικών συνηθιών. Στην Ισπανία ή στις χώρες μάλλον που δεν χρησιμοποιείται ευρέως το ελαιόλαδο, που χρησιμοποιείται μόνο εξαιρετικά, όντω εκεί οι τιμές είναι στα ύψη. Αυτό το αποφασίζουν όμως τα σούπερ μάρκετ. Τις τιμές δεν τις ε, καθορίζουν ε, οι κλάδοι, η, η διάρθρωσή τους. Πραγματικά ε, εγώ το πιστεύω. Δεν ξέρω τι λένε οι παραγωγοί της Ίστρια και σίγουρα είναι εξαιρετικό το ελαιόλαδο της Ίστριας. Είναι ιδιαίτερα ποιοτικό, άριστο, αλλά νομίζω ότι η προσθήκη μιας νέας κατηγορίας δεν θα βοηθήσει σε τίποτα και για τους παραγωγούς και για τον κλάδο δεν νομίζω ότι είναι θετικό το να προσθέσουμε μια νέα κατηγορία. Για την ε, θέση εμπορία ή για το σούπερ μάρκετ ίσως βολέψει μια νέα κατηγορία, αλλά για τους παραγωγούς όχι. Και μάλιστα είναι κατά της προσθήκης μιας κατηγορίας που θα επιφέρει μεγαλύτερη ακόμη σύγχυση. Γιατί την προσθεμένη αξία ε, την ε, φέρνει στο ελαιόλαδο ο χυμό του ελαιόλαδου που θα πρέπει να είναι χωρίς χημικά, χωρίς μεταποίηση, χωρίς αφινάρισμα. Αυτή είναι η προστιθέμενη αξία του ελαιόλαδου. Και νομίζω ότι είναι σαφές. Σέβομαι τη γνώμη σας κύριε Γιακόφτσιτς, αλλά συμφωνώ με τη συνάδελφο Εράς Γκαρσία. Για μας, τους Ισπανούς, ε, δεν θεωρούμε ότι μια νέα κατηγορία θα ωφελεί στον κλάδο. Αντίθετα θα επιτείνει τη σύγχυση και μπορεί να ευνοήσει τα σούπερ μάρκετ ίσως, αλλά όχι τους παραγωγούς που είδε ζήτησαν και θέλουν ξεκάθαρα πράγματα. Ε, παρθένο ελαιόλαδο, εξαιρετικό παρθένο ή ραφιναρισμένο μετά από χημική επεξεργασία δηλαδή. Είναι σαφείς οι κατηγορίες και δεν χρειάζονται περισσότερες. Δεν έχουμε ε, ε, άλλο ελαιόλαδο. Τα υπόλοιπα είναι προκαθορισμένα. Έχουμε το πυρηνέλο για παράδειγμα, αλλά υπάρχει ξεχωριστή κατηγορία. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Εράνς. Δεν είναι αυτό το αίτημα των παραγωγών, τουλάχιστον των παραγωγών στην Ισπανία. Σας ευχαριστώ κύριε Ντές που με αφήσετε να λάβω πρώτα το λόγο. ο κύριο Δες από τις ε, Ελαιώνες της Βαβαρίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που μίλησαν οι δύο Ισπανοί συνάδελφοι γιατί ήμουν πολύ θετικός να στην πρόταση του κυρίου Γεύκοβιτς. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα... αν υπάρχει ένα premium νομίζω θα μπορούν να κερδίσουν και περισσότερα η παραγωγή. Βεβαίως δεν είμαι ειδικό, αλλά κοιτώντα βεβαίως ε, τη, την γαλακτοπαραγωγή τη δική μου έχουμε ένα δισεκατομμύριο τζίρο και βεβαίως έχουμε και μια μάρκα premium που έχουμε 60 εκατομμύρια ε, τζίρο με πολύ ακριβότερη βεβαίω τιμή από τα στάνταρ προϊόντα. Οπότε μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση. Τώρα για την ερώτηση συναδελφοί του Κάστρο. Ήμασταν στην ε, Νότια Ιταλία και βεβαίως όταν βλέπει κανείς μια ελιά που υπάρχει 2.000 χρόνια τον πιάνει ιδέως ε, και πραγματικά νομίζω ότι από αυτά τα πολύ αρχαία δέντρα μπορούν, ε, μπορούμε να πούμε ότι το λάδι που βγαίνει θα μπορεί να πωλείται πάρα πολύ ακριβά γιατί βεβαίως κοστίζει και 50 ευρώ η φροντίδα του δέντρου το έτος, ενώ ένα πιο νέο δέντρο κοστίζει 5 ευρώ το έτος να το φροντίσουμε. Οπότε θα μπορούν νομίζω να πουλήσουν πιο ακριβά το λάδι του για να διατηρήσουν και αυτά τα, τα παλιά δέντρα. Οπότε θεωρώ πως είναι πολύ λογική η πρόταση του συναδέλφου Γιάκοφτσιτς αλλά νομίζω αυτά τα ξέρουν καλύτερα οι συνάδελφοι από τις ε, χώρες που παράγουν ηλιέ. Παρά την κλιματική αλλαγή ακόμα στη Βαβαρία δεν έχουμε ηλιέ. Okay, ale szczegóły 5 Ναι, αλλά οι διαφορές από 5 με 500 ευρώ μιλούν από μόνες τους. Ο κύριος φέραν. Ο Φεράντ. Ο κύριος Φερά. Oui. Ναι, φερό όπως ο στρατάρχης. Πρόεδρε, είναι πολύ σημαντικό το θέμα της, του ελαιολάδου. Έχουμε μείνει όμοιροι μια σειρά εξαγωγών αδασμολόγητων. Συμφωνώ με τις προτάσεις για τους ελέγχους, για την ποιότητα, για τις προδιαγραφές. Αλλά υπάρχει ένα τεράστιο θέμα εδώ που πρέπει να μας απασχολήσει σχέση με το ελαιόλαδο. Πρόληψη των ε, απατών και της παραποίησης της περιοχής προελεύσεως. Εάν δεν πάει κανείς να αγοράσει στον παραγωγό, βρίσκεται ενώπιον διαφόρων χαρμανίων από πολλέ χώρε, εταιρείε κτλ. που κάνουν ακριβώ αυτά τα χαρμάνια και που ω εκ τούτου εξαπατούν τον παραγωγό για, ε, στο θέμα τη προέλευση. Άρα χρειάζεται και η ποιότητα, όπω είπαμε, αλλά και η βεβαιότητα ότι το προϊόν είναι προϊόν προελεύσεω συγκεκριμένη. Σα ευχαριστώ. Δεν ζήτησε άλλο κανεί το λόγο από την ομίγυρη. Α, ο κύριος Δες, πάλι. Äh, Όλα αυτά ε, ε, ξαναπήρα τον λόγο. Μπορεί να μην είμαι παραγωγός, αλλά είμαι καταναλωτής ε, βεβαίως. ελαιολάδου. έκτιμω το προϊόν, ειδικά όταν πήγα στην Ιταλία. Μήπως θα μπορούσαμε να έχουμε μια αγορά premium από αυτά τα αρχαία δέντρα με κάποια εγγύηση όμως όπως μόλις ε, ακούστηκε γιατί εγώ θα πλήρωνα ευχαρίστως ε, παραπάνω για να συνεισφέρω στην διατήρηση αυτών των ε, δέντρων που έχουν ηλικία χιλιετιών. Αλλά να υπάρχει μια πιστοποίηση πράγματι, παραδείγματος χάρη για την ηλικία των δέντρων. Ε, Φαντάζομαι στην Ισπανία θα μπορούσαμε να βρούμε τέτοιες ελιές ε, και να πληρώνουμε και 100 ευρώ για τέτοιες ελιές που προέρχονται από υπεραιωνόβια ελαιόδεντρα. Δεκάστρο. Θα ήθελα να διευκρινίσω μία πτυχή και δεν είχα λάβει το λόγο πιο πριν γιατί η Κλάρα και η Αράνς Καρσία ήδη είχαν ξεκαθαρίσει το θέμα αυτό. Αλλά Άλμπερτ πρέπει να διευκρινίσουμε το εξή. Άλλο είναι η διεθνή ταξινόμηση γνωστή σε όλους μας που ορίζει το αγνό παρθένο, απλό παρθένο και ούτω καθεξής ελαιόλαδο. Αυτό είναι γνωστό και για τον παραγωγό και για τον καταναλωτή. Αλλά είναι κάτι διαφορετικό το να μιλήσουμε για τις ε, εθελοντικές και ιδιωτικές ίσως δυνατότητες που έχει ένας ε, παραγωγός να ταυτοποιήσει το προϊόν του, όπως η παραγωγή της πουλιας, που βάζουν ένα ειδικό σήμα όταν πρόκειται για ε, εκατονταετής ε, για αιωνόβιες ελιές. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι μια, ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό και θέλω να το διευκρινίσω συμφωνώντας με την ε, Κλάρα και την Εράντς ότι Άλλο πράγμα είναι η διεθνής ταξινόμηση, αλλά επιπλέον αυτή θα μπορούσαμε να έχουμε είτε ιδιωτικό σήμα είτε και συλλογικά σήματα που θα έδιναν χαρακτηριστικά μια μιας σε μια συγκεκριμένη περιοχή, ενδεχομένω η ζώνη. Και επίσης πέραν αυτού οι ονομασίες γεωγραφικής προελεύσεως που ξέρετε ότι μας ε, έχουν απασχολήσει και έχουμε δώσει τη δυνατότητα να βάλουμε πέραν της γεωγραφικής προελεύσεως και το χαρακτηριστικό φερρυπίν Ορεινή παραγωγής, για το τυρί. Ε, το ίδιο θα μπορούσαμε ίσως να συζητήσουμε και για την ελιά, αν και θα καταστούσε τα πράγματα αρκετά περίπλοκα και ίσως να οδηγούσε σε σύγχυση. Μάλιστα. Θα ζητήσουμε τώρα από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν θέλει να λάβει το λόγο. Ο κύριος Χάπς. Θέλετε το λόγο, κύριε Χάπς. Ναι, από ό,τι φαίνεται. Παρακαλώ, έχετε το λόγο, κύριε Διευθυντά. Thank uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και κύριε Γιάκοβτσιτς ε, για την έκθεση αυτή. Χαιρόμαστε οπωσδήποτε που εγκρίνεται την την συμφωνία με το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου και ήταν δύσκολη δουλειά για εμάς, ε, ήταν μια διεθνής συμφωνία και η νέα συμφωνία είναι ένα μεγάλο επίτευγμα γιατί ακριβώς ε, καθορίζει στο διεθνές επίπεδο τα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελαιών. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την στήριξή σας ε, και θα τόνιζα ότι χαιρόμαστε που μπορούμε να ξεκινήσουμε ε, με την προσωρινή εφαρμογή της ε, συμφωνίας αυτής που ισχύει από πρώτης πρώτου και ίσως ε, από του χρόνου να έχουμε οριστική εφαρμογή. Αυτό το οποίο επίσης θα ήθελα να αναφέρω είναι το θέμα ενός, μιας άλλης επιπρόσθετης προδιαγραφής ποιότητας είναι πολύ δύσκολο. Επί της αρχής έχουμε τις τρεις ε, κατηγορίες, εξαιρετικό παρθένο, παρθένο και λαμπάντε, ε, που πολλούνται εντός της Ένωσης ε, και διεθνώς ως διεθνώς αναγνωρισμένες βαθμίδες ποιότητας και ξέρετε ότι αυτές είναι τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στα διάφορα παραρτήματα και στην ε, σχετική βεβαίως ε, συμφωνία. Έτσι έχουμε οργανώσει τις ποιοτικές μας προδιαγραφές ε, στην Ευρώπη και διεθνώς, γιατί υπάρχει και διεθνές εμπόριο, όχι μόνο εξάγουμε εξαιρετικά παρθένο, ελαιόλαδο, στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά εισάγουμε κιόλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίω το να μπει άλλη μια προδιαγραφή είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει στο πλαίσιο του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου και οπωσδήποτε αυτό θα χρειαζόταν και την, εγγύηση, και την έγκριση με συγχωρείτε, άλλων εταίρων. Δεν μπορεί να αποκλειστεί, θα το κάνουμε εάν είναι αναγκαίο αλλά για μένα προσωπικά και για πολλούς ε, παραδοσιακούς παραγωγούς θα έλεγα ότι έχουμε και άλλα μέσα για να προστατεύσουμε το ελαιόλαδο ποιότητος πέρα από το εξαιρετικό παρθένο κυρίως και ιδιαίτερως μέσω των 120 pop και των ε, γεωγραφικών, προστατευμένων γεωγραφικών ενδείξεων. Επίσης υπάρχει δυνατότητα και οι καταναλωτές να ξέρουν ότι δεν είναι μείγμα διαφόρων προελεύσεων ε, από, διάφορους, ε, από διάφορα μέρη ή διάφορες ποιότητες. Για απαντήσω στον κύριο Ντέστορα τα παλιά δέντρα είναι εντάξει, πάρα πολύ ωραία στην όψη, αλλά δεν είναι εγγύηση υψηλής ποιότητας λαδιού. Να είναι βεβαίως κάτι που θα χρησιμοποιηθεί για το μάρκετινγκ, αλλά η έλεγχη ποιότητα είναι τεχνική έλεγχη και πρέπει να σεβόμαστε τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και τις ε, χημικές αναλύσεις. Αυτά για εμάς είναι η ένδειξη της ποιότητας. Επίσης ο εισηγητής ε, αναφέρθηκε στο πώς θα οργανωθεί στο μέλλον ο καταμερισμός εργασίας μεταξύ Συμβουλίου και Κομισιόν για τις Διεθνείς ε, Συμφωνίες. Αυτό δεν είναι κάτι ε, συγκεκριμένα για το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου και πρέπει να παραδεχτώ ότι ακόμα συζητάμε με το Συμβούλιο και είναι βεβαίως και ένα θέμα μεταξύ των δύο νομικών υπηρεσιών. Προσωπικά είμαι αισιόδοξο ότι θα καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα που θα λύσει το πρόβλημα έτσι ώστε να μπορούμε να είμαστε επιχειρησιακοί, ειδικά στο Συμβούλιο Ελαιολάδου, γιατί ε, είναι ένας από τους πιο ζωντανούς και σημαντικούς ε, διεθνείς οργανισμούς για να προωθήσουμε ένα συγκεκριμένο προϊόν στον κόσμο και βεβαίως να εγγυόμαστε και την ποιότητα για τους καταναλωτές. Σας, ευχαριστούμε. Ο εισηγητής μας, ο κύριος Γιακόφτσης τώρα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Χαίρομαι που κανείς δεν αντιτάχθηκε στο να δώσουμε το πράσινο φως για την ε, σύναψη και οριστικοποίηση αυτής ε, της Διεθνούς Συμφωνίας για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές από το 2015. Χαίρομαι που κάνετε δεκτή τη γνωμοδότησή μου. Ε, νομικά μόνο αυτό δικαιούμαστε, να δώσουμε τη συνένεσή μας ή να αντιταχθούμε. Αλλά χαίρομαι γιατί είχαμε πραγματικά πολύ καρποφόρα συζήτηση. Αυτό περίμενα άλλωστε επικοδομητική συζήτηση. Εγώ ήθελα απλώ να σας πω ότι μετά από συζήτηση που είχα σε κάποιες ε, χώρε και με κάποιους παραγωγούς, γιατί πήγα και στην Κόπα Κοζέκα και εκεί συζήτησα με τους παραγωγούς και στην Κόπα Κοζέκα ε, γίνονται συζητήσεις ε, διαφόρων προτάσεων. Νομίζω ότι είναι σκόπιμο να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία συζήτηση και διαλόγου με ώστε κάποια μέρα και με κάποιο άλλο τρόπο να προστατεύουμε την προέλευση, γιατί όπως ξέρετε το καλύτερο ελαιόλαδο σχεδόν αποκλειστικά παράγεται στο επικράτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο από Ευρωπαίους δηλαδή παραγωγούς ουσιαστικά. Και πολύ συχνά έχουν το ελαιόλαδό τους και το αποκαλούν εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, αλλά λένε ότι έχουν προβλήματα με την ποιότητα πολλές φορές. Και πολλές φορές φτάνουν στι αγορές μας ελαιόλαδα από χώρες νοτίους Μεσογείου που είναι χειρότερης ποιότητας. Και αυτό μερικές φορές το στηρίζουν τα σούπερ μάρκετ και... ή το ανέχονται. Ε, είμαστε η το ανεχονται παραγωγή ελαιολάδου στον κόσμο. Οι Ευρωπαίοι παραγωγοί ελαιολάδου είναι οι καλύτεροι. Παράγουν αρίστης ποιότητα ελαιόλαδο, γι' αυτό και καλό θα είναι να μένουν ικανοποιημένοι και οι παραγωγοί και οι καταναλωτές μας. Δεν συμφωνώ με τις συναδέλφους ότι με τον προσδιορισμό μιας νέας κατηγορίας θα επιτείνουμε τη σύγχυση στου καταναλωτές. Εδώ διαφωνούμε. Πολύ μεγαλύτερη σύγχυση υπάρχει όταν ε, με, την, ε, με πολύ διαφορετικές τιμές ε, τα ίδια ποιότητα, το εξαιρετικά παρθένο, γιατί σας είπα πόσο μεγάλη είναι η ψαλίδα των τιμών, από 4 ευρώ το κιλό το λίτρο μέχρι 30. Και τότε πραγματικά μπερδεύονται οι καταναλωτές. Πώς είναι δυνατό για την ίδια ποιότητα ελαιολάδου να είναι τόσο διαφορετικές οι τιμές. Γι' αυτό έχουμε κατά τη γνώμη μου πρόβλημα. γι' αυτό πρότεινα το, το σχετικό ζήτημα για να γίνει συζήτηση. Και χαίρομαι γιατί το σημαντικότερο είναι ειλικρινά και έντοιμα να μιλούμε μεταξύ μα, ώστε καθένα από εμά να προστατεύει και τα εθνικά του συμφέροντα και τα συμφέροντα των εθνικών παραγωγών, αλλά να ξεκινήσουμε μια διαδικασία, γιατί επαναλαμβάνω το 15% το, του αερί τη ποιότητα ελαιολάδου στον κόσμο παράγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή είναι ε, ένας υπολογισμός, αυτός είναι ένας υπολογισμός που έκαναν Ιταλοί συνάδελφοι. Πιστεύω θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη και να βοηθήσουμε τους παραγωγούς μας και τους καταναλωτές μας φυσικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε εισηγητά. Όπως είπε και ο εισηγητής, απλώς πρέπει να δώσουμε τη συνένεση, να πούμε ναι ή όχι για τη σύναψη της συμφωνίας, την οριστικοποίηση της. Και έχετε και μία προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών, πολύ σύντομη. Ουσιαστικά πρέπει να πούμε ναι ή όχι στη σύναψη της συμφωνίας για το ελαιόλαδο και αρμόδια κατ' ουσίαν είναι η Επιτροπή Διεθνούς Εμπόριου, η Επιτροπή ΙΝΤΑ όπως είπαμε. Η έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης θα γίνει στην επόμενη μας συνεδρίαση και η αρμόδια κατ' ουσίαν Επιτροπή Ίντα θα ψηφίσει στις 4 Δεκεμβρίου. Ωραία, ολοκληρώσαμε αυτό το θέμα, το 5, και περνάμε στη συζήτηση για τις επιπτώσεις του Brexit. Καλό θα ήταν για να προετοιμάσουμε τις παρουσιάσεις, να κάνουμε μία σύντομη διακοπή ένα πεντάλεπτο διάλειμμα. Πέντε λεπτά μόνο όμως, όχι παραπάνω. Πεντάλεπτο διάλειμμα παρακαλώ. Συνάδελφοι, έχουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, γι' αυτό και θα αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο στα επιμέρους ζητήματα. Έχουμε τρεις εκθέσεις, όπως ξέρετε, τρεις μελέτες που έγιναν, που αφορούν τα θεσμικά, δημοσιονομικά και θεσμικά ζητήματα τις θεσμικές, δημοσιονομικές και εμπορικές πτυχές. Ε, πρόκειται για μελέτες που ζητήθηκε από την Επιτροπή Γεωργίας και διεξάγονται από το Τμήμα Πολιτικών Β. Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα των επιπτώσεων του Brexit στο μέτρο που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσει, αλλά που δεν έχουν παρουσιάσει μέχρι στιγμή ιδιαίτερη πρόοδο. Και σε αυτό το καιρό τη βεβαιότητα, η Επιτροπή Γεωργία και το Τμήμα Πολιτικών Β οργάνωσαν αυτό το εργαστήριο, το σεμινάριο με τίτλο Συνέπειε του Brexit για τον ε, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Κλάδο και την Κοινή Γεωργική Πολιτική». Με ε, συμβολή και συνεισφορά κορυφαίων Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων. Θα ασχοληθούμε με τι βασικέ δημοσιονομικέ, εμπορικέ και θεσμικές πτυχές ε, που σχετίζονται με το Brexit. Και έχουμε τρία θέματα στο εργαστηριό μας. Καταρχήν το πιθανό αντίκτυπο του Brexit ε, για τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό και ιδιαίτερα για τη χρηματοδότηση ΚΑΠ. Εδώ θα έχουμε δύο εμπειρογνώμονες, την κυρία Ευλαλία Ρούμπιο και τον κύριο Γιώργ Χάς από το Ίδρυμα Jacques Delors και την Ευρώπη μας. Το δεύτερο τμήμα, η δεύτερη θεματική ενότητα αφορά το γεωργικό εμπόριο Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου και την κατάσταση πιθανές συνέπειες από το Brexit. Ε, θα έχουμε εδώ την κυρία Σεσίλια Μπελόρα, ομιλήτρια, και τον κύριο Ζαν Φουρέ από το ε, Κέντρο Διεθνών Σπουδών και Οικονομικής Διαχείρισης του Παρισιού. Και το τρίτο θέμα θα είναι οι πιθανές ε, μεταβατικές ρυθμίσεις για τη γεωργία υπό το φως των μελλοντικών σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου. Θεσμικές πτυχές δηλαδή, θα μας εξηγήσει ο κύριος Άλαν Μάθιος, γνώριμος της Επιτροπής μας, επίτιμος καθηγητής του Trinity College του Δουβλίνου. Χαιρόμαστε ιδιαίτερως και για την παρουσία του. Για κάθε θέμα οι ομιλητές θα έχουν 20 λεπτά στη διάθεσή τους, θα ακολουθήσει σε ερωτήσεων. Αλλά ερωτήσεων, το τονίζω παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι γιατί η συζήτηση θα γίνει μετά την ολοκλήρωση και των τριών παρουσιάσεων. Μετά την κάθε επιμέρους παρουσίαση θα γίνουν μόνο ερωτήσεις, θα απαντά ο εμπειρογνώμονας, ακολουθεί δεύτερος εμπειρογνώμονας, δεύτερο θέμα, παρουσίαση και μετά ερωτήσεις, τρίτο θέμα το ίδιο και στο τέλος θα γίνει συνολική συζήτηση εφόλης της ύλης, των τριών θεμάτων δηλαδή. Έχουμε αρκετό χρόνο για αυτό το σεμινάριο και παρακαλώ περάσουμε στους καλεσμένους μας Ξεκινάμε με το πρώτο θέμα, τις δημοσιονομικές πτυχές. Παρακαλώ, η κυρία ρούμπι. Thank you Thank you very much. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε το λόγο και που μας προσκαλείτε σε αυτό το εργαστήρι. Ε, καθήκον μας ήταν η ανάλυση των δημοσιονομικών συνεπειών του Brexit για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και ιδιαίτερα στις δαπάνες της κοινή γεωργικής πολιτικής. Αυτή είναι η δομή λοιπόν ε, της παρουσίασης λίγο πολύ και της μελέτης. Είχε να κάνει με την ανάλυση της κατάστασης και ιδιαίτερα των συνεπειών των διαπραγματεύσεων πώς μπορεί να επηρεάσουν το τρέχον δημοσιονομικό αλλά και το μελλοντικό δημοσιονομικό πλαίσιο και βέβαια συγκεκριμένα με την ε, ε, συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στον προπολογισμό. Και στη, το δεύτερο κομμάτι που θα παρουσιάσει ο συνάδελφο είναι συγκεκριμένα οι συνέπειε τη δαπάνη τη ΚΑΠ. Θα κλείσουμε δε με ε, συμπεράσματα και συστάσει. Πριν περάσω στα δύο ζητήματα των επιπτώσεων, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι θα προκύψουν διάφορες συνέπειες του Brexit για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, πέραν των δύο που ανέφερα το κόστος και το διαρθρωτικό, διαρθρωτικές συνέπειες. Μπορεί να έχουμε σημαντικές ε, συνέπειες και στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η ιδέα απουσία του Ηνωμένου Βασιλείου από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων μπορεί να αλλάξει και τη δυναμική στο τραπέζι του των διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο. Επίσης, θα ενισχυθεί ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός σε σχετικούς όρους, σε όρους ΑΕΠ, Γιατί ακόμη και αν κάνουμε την προσαρμογή του κενού του Brexit, δηλαδή των συνεπειών της αποχώρησης, με την αύξηση των δαπανών παραμένει το αποτέλεσμα ενός ευρωπαϊκού προπολογισμού μεγαλύτερου σε πραγματικού όρου και παρά την επιστροφή τη Βρετανική. Γιατί ξέρετε ότι αυτό έχει πολλές φορές ε, σημειωθεί ότι δεν θα πρέπει να αυξηθεί κατά 1% το ΑΕΠ. Όχι, αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Και βεβαίως, επιπλέον, συνέπειες ως προς τους ιδίους πόρους, γιατί θα αλλάξουν τα συστήματα διορθώσεων με την ε, αποχώρηση από το σύστημα της Ευρωπαϊκής Βρετανικής Επιστροφής. Άρα μπορεί να οδηγηθούμε σε διαφορετικά συμπεράσματα σχέση με την μεταρρύθμιση συστήματος των ιδίων πόρων. Ε, ξέρετε, ο λογαριασμό του Brexit, όπω λέγεται, Brexit Bill, έχει να κάνει με το κόστο των διαπραγματεύσεων. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πληρώσει το δικό τη μερίδιο από τι οικονομικέ δεσμεύσει που έχουν από κοινού αναλυφθεί από πλευρά των κρατών μελών, όσο ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο μέλο Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, έχουμε να κάνουμε την προσαρμογή στο Brexit και όχι με μελλοντικέ πληρωμέ ή το κόστο μια μελλοντική εταιρική σχέση. Όταν ετοιμάζαμε το έγγραφο που ήμασταν ακόμη στη φάση την πρώτη των διαπραγματεύσεων του Brexit, η οποία όπως θα γνωρίζετε δεν έχει τελειώσει, και βέβαια η διαθέτηση των οικονομικών έχει παραμείνει το κύριο αγκάθι στην πρώτη αυτή φάση, γιατί υπάρχει ακόμα σημαντική απόκληση στι θέσει μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο προ τα ποσά, αλλά και τη φύση και τα νομικά ζητήματα των διεκδικήσεων και απαιτήσεων αυτών. Τώρα έχουμε ένα ευρωπαϊκό έγγραφο αρκετά λεπτομερέ του Ιουνίου του 2016, με ένα κατάλογο των δημοσιονομικών υποχρεώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, όπω τι βλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οφειλόμενα δηλαδή από πλευράς Ηνωμένου Βασιλείου και πώς θα πρέπει να ε, καταβληθούν χωρίς συγκεκριμένα ποσά ε, στο έγγραφο, ωστόσο με κάποιους υπολογισμούς βλέπουμε ότι θα φτάσει κάπου στα 55 με 75 δισεκατομμύρια. Και το άλλο στοιχείο είναι η σαφέστερη μέχρι τώρα δήλωση της Τερέζα Μέη και, της, και η ε, δέσμευσή της στην ομιλία της στη Φλωρεντία του Σεπτέμβριου του 2016. Λέει ομιλήτρια ε, ότι δεν θα ε, αφήσει εκτεθειμένο κανένα κράτη και έτσι θα καλύψει τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις του 2020, δηλαδή περί τα 20 δις είναι κάτι το οποίο συζητεί πολύ ο Τίτο, ότι υπάρχουν αποκλήσει μεταξύ των δύο ποσών, των ποσών που παρουσιάζουν οι δύο πλευρέ. Αλλά βέβαια υπάρχουν, όπω είπα, και άλλα ζητήματα, νομικά και πολιτικά, οι σχετικέ απαιτήσει. Πρώτον, για το φύση του λογαριασμού αυτού. Και υπήρξαν κάποιες πρόσφατες αναφορές στον τύπο για αλλαγές ίσως, θα τις είδατε κι εσείς, Φαίνεται δηλαδή να είναι διατεθειμένο το Ηνωμένο Βασίλειο τώρα να αυξήσει τα ποσά στο λογαριασμό, αλλά πάντα παραμένουν οι διαφωνίες ως προς το ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να συνδυάσει την καταβολή των ποσών με την φάση, με την φύση των μεταβατικών ρυθμίσεων γιατί βέβαια θα είναι πολύ πιο εύκολο για το Ηνωμένο Βασίλειο να ε, παρουσιάσει στην κοινή του γνώμη αυτές τις πληρωμές ως ε, κομμάτι των μεταβατικών διατάξεων, αλλά ταυτόχρονα από την πλευρά Ευρωπαϊκής θα πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα ώστε την ε, συμφωνία αυτή να μην την συνδυάσουμε με μια μεταβατική υποτιθέμενη συμφωνία, διότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί σε δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων. Ε, υποχρεώσεις. Ένας κατάλογος που θα δείτε στον, ε, στις διαφάνειές μας, κατάλογος των υποχρεώσεων που αναφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που περιλαμβάνει στο λογαριασμό. Ε, κάτι που είχε στηθεί αρκετά ήταν οι συντάξει, αλλά δεν το μεγαλύτερο ποσό αυτό. Το μεγαλύτερο ποσό είναι αυτό που έχει να κάνει με τις δαπάνες και ε, υποχρεώσεις δαπανών που σχετίζονται με το τρέχον δημοσιονομικό πλαίσιο. αμφισβήτηση υπάρχει ως προς το αν θα πρέπει όλες τις ε, υποχρεώσεις που σχετίζονται με το πολίτες πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τις καταβάλει το Ηνωμένο Βασίλειο ή αν θα πρέπει να περιοριστεί μόνο στο προϋπολογισμό. Γιατί υπάρχει βέβαια ο ετήσιος προϋπολογισμός, αλλά ξέρετε ότι υπάρχουν και τα περίφημα αράλτα, υπόλοιπα προς ρευστοποίηση Οπότε αν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε το 2019 θα έχει να πληρώσει τα ράλη του 2019, αλλά υπάρχει και αμφισβήτηση για το αν το Ηνωμένο Βασίλειο έχει να πληρώσει όλες τις ε, αναλήψεις υποχρεώσεων ε, που έχουν ε, συμπεριληφθεί στο τρέχον στο νομικό πλαίσιο, αλλά όχι στον αιτήσιο προπολογισμό. Ενώ κάποιοι λένε ότι θα πρέπει να αναγνωριστούν οι απαιτήσει για τους ενοποιημένου ευρωπαϊκούς λογαριασμούς, όχι όλες δηλαδή οι δαπάνε, αλλά οι αναλήψεις υποχρεώσεων οι και φαίνεται ότι η Τερέσα Μέη στην ομιλία της της ε, Φλωρεντίας ε, λίγο πολύ το δέχεται. Ένα άλλο ζήτημα είναι οι λοιπές απαιτήσει. ενδεχόμενες απαιτήσει, όπου θα πρέπει το Ηνωμένο Βασίλειο να καταβάλει ένα ποσό ε, αρχικό από απαιτήσει που ενδεχομένως να ε, υλοποιηθούν στο μέλλον. Άρα καταλαβαίνετε από αυτά που σας λέω ότι μπορεί να είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση ανάλογα με το αν θα πληρώσετε τα υπόλοιπα προς ε, ρευστοποίηση του Ηνωμένο Βασίλειο ή όχι. Και βέβαια η συμμετοχή του στον προπολογισμό για το 19 και το 20 ε, αμφισβητείται εάν δεν εγγραφεί στον ε, τίσιο προϋπολογισμό για το 19 και το 20 ε, η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά περιοριστεί μόνο στους ενοποιημένους λογαριασμούς, τότε αμφισβητείτε αν θα καλυφθούν όλες οι, δαπάνε, δαπάνες ε, των διαρθρωτικών ταμείων, γιατί βέβαια αυτό περιλαμβάνεται σε ένα βαθμό, ε, μάλλον αυτές περιλαμβάνονται σε ένα βαθμό στις αναπαιδευμένους λογαριασμούς, αλλά όχι του ε, Ευρωπαϊκού Ταμείου ε, το, του ΕΚΤΠΑ. Το ίδιο υπάρχει περίπτωση να δεχθούν να πληρώσουν τις αιτήσιες, την ετήσια συμβολή, αλλά όχι τα εκκρεμή για το 2020 ραλ. Και άρα παραμένουν οι δαπάνες της ΚΑΠ για το 19 και το 20, αλλά ε, θα είναι πολύ πιο δύσκολες οι διαπραγματεύσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο το 27 για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο δηλαδή. Διαρθρωτικές συνέπειες ο μόνιμος αντίκτυπος της αποχώρησης, του έλλειψης του Ηνωμένου Βασιλείου. Βέβαια ξέρουμε ότι από τώρα ένα χρόνο στον άλλο μπορεί να αλλάξει. Ε, έχουμε υπολογισμούς του 14 με 16, έχουμε ένα ποσό περί τα 10 δις ως απώλεια για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Εδώ θεωρούμε ότι το Brexit θα έχει μορφή σκληρή, δηλαδή χωρίς συμφωνία για μετά το 2020. Αυτό είναι ένα από τα σενάρια, 10 ε, δις λοιπόν το χρόνο και πώς μπορούμε να το καλύψουμε το ποσό αυτό, πώς μπορούμε να προσαρμοστούμε. Έχουμε διαφορετικά σενάρια, έχουμε αναλα... αναλύσει διάφορα σενάρια προσαρμογής με την αύξηση των συνεισφορών των κρατών μελών ένα άλλο έχει να κάνει με μείωση των δαπανών. Αλλά κάναμε και ένα σενάριο με υπόθεση τι θα γίνει αν δεν υπάρξει συμφωνία για τις διαπραγματεύσεις πολίτου του δημοσιονομικού πλαισίου. Ε, επίσης υπάρχουν άλλες δυνατότητες ε, σενάριων πιο περίπλοκων που δεν έχουμε αναλύσει στην ε, τρέχουσα παρουσίαση. Αλλά πολύ ευχαριστώ να σας απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας. Στο πρώτο σενάριο λοιπόν βλέπετε το ποσό. Εάν ζητηθεί να αυξηθούν οι συνεισφορές των κρατών μελών, στο πάνω μέρος της γραφικής παράστασης βλέπετε ποσοστό εθνικών συνεισφορών, ποσοστό αύξηση των εθνικών συνεισφορών, ενώ στο κάτω μέρος βλέπετε τα ε, καθαρά ποσά. Και βέβαια η χώρες οι οποίες συνεισφέρουν τα μάλα στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό θα έχουν τη μεγαλύτερη επιβάρυνση σε πραγματικά ε, ποσά, αλλά κυρίως αυτές οι οποίες έχουν επιστροφή θα έχουν αναλογικά τη μεγαλύτερη επιβάρυνση. Από την κατάργηση του της διόρθωσης για το Ηνωμένο Βασίλειο της επιστροφής πάβουν και οι αντίστοιχες διορθώσεις για τη Γερμανία, τις κάτω χώρες και τη Σουηδία που θα πληγούν περισσότερο αναλογικά από το πρώτο αυτό σενάριο. Στο εσενάριο 2 κοιτάμε να δούμε τι θα γίνει εάν μειωθούν οι δαπάνες. Και περιγράφουμε τις δυσκολίες ανάμεσα του σενάριου. 10 δισεκατομμύρια σε έναν προϋπολογισμό των 130 είναι πολλά χρήματα, είναι μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού και προσπαθούμε να περιγράψουμε τρόπους για περιορισμό των δαπανών σε διάφορα προγράμματα που όπως βλέπετε σημαίνει 20% στις τρέχουσες ε, δαπάνες για τη συνοχή και συνολικά όλο τον προπολογισμό του Ρωστα 2000, ε, περικοπή σε πάρα πολλά άλλα προγράμματα, στην ΚΑΠ κτλ. Ε, πάρα πολύ μεγάλα ποσά, δηλαδή αν χρειαστεί να γίνει ε, προσαρμογή στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, μόνο μέσω των δαπανών στον του... μόνο περιορισμού των δαπανών στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Και το τρίτο σενάριο είναι τι γίνεται αν δεν προκύψει συμφωνία. Δύο σενάρια εδώ πέρα, είτε θα πρέπει να γίνει προσαρμογή πριν από το 2020, στο Brexit. Δηλαδή υπολογίζουμε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία Brexit. Φεύγει το Ηνωμένο Βασιλείο 2019 με συμφωνία να καταβάλει τις καθαρές εισφορές στο 2020, που πάλι δεν είναι σαφές ότι θα συμβεί. Έχουμε τον τρέχοντα κανονισμό του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, που όμως δεν προβλέπει συγκεκριμένο τι μπορεί να γίνει, μόνο ότι πρέπει να προσαρμόσετε σε αλλαγές συνθήκης ε, το πουδουπού Πιο συγκεκριμένους όμως όρους δεν, δεν έχουμε στην νομοθεσία αυτή. Και το άλλο θα είναι αν δεν υπάρχει κάλυψη μετά το 2019. Άρα τα όρια του, των δαπανών του τρέχοντος MFF για, το, για την περίοδο 19-20 το τελευταίο έτος, δηλαδή μετά την αποχώρηση του, των Βρετανών, θα πρέπει να διατηρηθούν ως επίπεδα δαπανών, αλλά πάλι παραμένουμε σε μια εκκρεμότητα γιατί δεν ξέρουμε νομικά τι ισχύει εάν έχουμε τόσο υψηλά ε, όρια δαπανών. Και αυτό θα επηρεάσει και τα κράτη καθαρούς ε, συνεισφέροντε αλλά και τους καθαρού αποδέκτες. Και ο συνάδελφος τρόπο να συνεχίσει. Να είμαστε πιο συγκεκριμένα τώρα. Τι σημαίνουν αυτά για την ε, γεωρική πολιτική, πώς μπορεί να προσαρμοστεί και τι σημαίνουν για τα κράτη-μέλη. Πρώτα απ' όλα Α δούμε μια ματιά στο status quo. Βλέπουμε εδώ πέρα τον ε, ισολογισμό της ε, κυνηγής γεωρικής πολιτικής σε εκατομμύρια ευρώ. Βλέπουμε πώ η ψαλίδα είναι μεγάλη, μεγαλύτερη και από την ψαλίδα Συνοχή. Υπάρχουν πέντε μεγάλε χώρε οι οποίε λαμβάνουν, Πολωνία τα περισσότερα, μετά Ελλάδα, Ρουμανία, Ισπανία, Ουγγαρία και από την άλλη έχουμε δύο μεγάλου καθαρού εισφορεί, ε, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Τι θα γίνει λοιπόν όταν φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο? Αφενό. Όπω είπε η συνάδελφο, υπάρχει ο λογαριασμό του Brexit που θα μπορούσε να επηρεάσει την κοινή γεωργική πολιτική και πριν το 2020. Δεν ξέρουμε τώρα πώς θα εξελιχθεί, μπορεί ναι, μπορεί όχι. Αλλά μετά το 2020 θα υπάρχει οπωσδήποτε κενό και κάποιος πρέπει να το γεμίσει. Το ερώτημα είναι πόσο θα πρέπει να συνεισφέρει η γεωργική πολιτική στο να κλείσει το κενό. Και δεν είναι σαφές. Βεβαίως, μπορούμε απλά να πάρουμε την βρετανική συνεισφορά και να πούμε αυτό είναι το κενό, δηλαδή 3 δισεκατομμύρια το έτος και να πούμε θα το χρεωθεί η ΚΑΠ. Αν όμως ε, λάβουμε υπόψη ότι το συνολικό χρηματοδοτικό κενό είναι 10 δισεκατομμύρια το έτος, τα μεγαλύτερα προγράμματα όπως η ΚΑΠ θα έχουν και το μεγαλύτερο έλλειμμα. Είναι πολιτικό όμως το ζήτημα και όσο κοιτάμε τις διάφορες επιλογές για το πώς μπορεί να προσαρμοστεί ε, Προπολογισμό της ΚΑΠ. Βλέπουμε το τι γίνεται στον τομέα τη γεωργικής πολιτική. Αυτά τα οποία θα σα παρουσιάσω είναι επιλογές, όχι προτάσεις. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσει να διατηρήσει τις ε, δαπάνες ε, της γεωργίας στο υφιστάμενο επίπεδο, οι εισφορέ πρέπει να αυξηθούν. Βλέπουμε τα αποτελέσματα. Κάτω βλέπετε τα απόλυτα ποσά σε εκατομμύρια ευρώ. Πάνω βλέπετε τον αντίκτυπο στις ε, κρατικές δαπάνες, πάντα σε σύγκριση με τα σημερινά. Οι μεγαλύτερε και πλούσιότερες χώρε επηρεάζονται περισσότερο γιατί οι επιπρόσθετε εισφορές βασίζονται στο ΑΕΠ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Όπως ε, είπε και η συνάδελφος, Αυστρία, η Γερμανία, Σουηδία και Ολλανδία επηρεάζονται περισσότερο γιατί χάνουν την επιστροφή, κάτι το οποίο είναι για αυτές κακό καλό για όλους τους υπόλοιπους. Ε, π.χ. Ολλανδία και Σουηδία θα έχουν τον ίδιο αντίκτυπο με την Ιταλία, παρά το ότι η Ιταλία έχει τρεις φορές μεγαλύτερη οικονομία. Είναι άδικο. Ναι, μπορεί να πει κανείς ότι είναι άδικο, αλλά μπορεί να πει ότι και το υφιστάμενο σύστημα τους δίνει κάποια άδικα πλέον εκτήματα αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι είναι δύσκολο πολιτικά το ζήτημα. Οι με καθαρείς φορείς ε, θα κληθούν να πληρώσουν περισσότερο, ενώ όσοι ε, λαμβάνουν ε, θα επηρεαστούν ελάχιστα. Εάν κόψουμε τις δαπάνες κατά τρία δις τώρα έχουμε κάποια μεικτά αποτελέσματα. Βλέπουμε ότι οι χώρες οι οποίες ε, λαμβάνουν αυτή τη στιγμή, Πολωνία και Ελλάδα, επηρεάζονται περισσότερο, αλλά βεβαίως επηρεάζονται και οι χώρες, οι καθαρές φορείς Γερμανία, Αυστρία κτλ. Πολιτικά αυτό δεν είναι κακό γιατί δεν θα υπάρξει ένα συνασπισμό ε, όσων λαμβάνουν ε, εναντίον όσων ε, πληρώνουν αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν ξέρουμε αν θα αρκούν τα 3 δισεκατομμύρια. Τι θα γίνει λοιπόν αν κόψουμε 10 δισεκατομμύρια. Ένα μάλλον ακραίο σενάριο ομολογουμένω, αλλά τονίζει κάποιε σημαντικέ αλλαγέ. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι αυτή τη φορά οι χώρε οι οποίε λαμβάνουν χάνουν πάρα πολλά και ειδικά σε σύγκριση με τις συνολικές δικές τους δαπάνες και η αλλαγή αυτή επηρεάζει ιδιαίτερα τις φτωχότερες χώρες όπως Ρουμανία, Βουλγαρία, Λιθουανία και βέβαια και αυτό είναι προβληματικό πολιτικά. Ταυτόχρονα οι καθαροί εισφορείς ε, κερδίζουν από αυτά τα σενάρια και μειώνονται οι ανισορροπίες στην ΚΑΠ. Αυτή τη διαφάνεια θα την περάσω, δεν έχουμε χρόνο. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι ε, το θέμα δεν είναι μόνο οι συνολικές περικοπές αλλά και οι λεπτομέρειες. Ανάλογα με το είδος των περικοπών μπορούμε να ε, προστατεύσουμε τα φτωχότερα κράτη-μέλη από τα χειρότερα. Συμπερασματικά λοιπόν. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει κάποιο τεχνικό τρόπο για να δούμε πόσο πρέπει να προσαρμοστεί η ΚΑΠ μετά τον Brexit. Μπορεί να μην επηρεαστεί καθόλου, μπορεί να είναι 3 δι, μπορεί να είναι 10 δι περικοπέ, μπορεί και περισσότερο. Δεύτερον, κανένα από τα σενάρια αυτά δεν είναι τέλειο. Βεβαίω υπάρχουν σαφή μειονεκτήματα. Αν μειώσουμε τις φορές, σημειώνουμε και τις ανισορροπίες. Αν κόψουμε κατά πολύ την ΚΑΠ, επηρεάζουμε πολύ τα φτωχότερα κράτη-μέλη. Ε, δεν υπάρχει λοιπόν κάποιο ανώδυνος τρόπος. Και τέλος, κάποιες συστάσεις. Θεωρούν πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι προσεκτική όσον αφορά την σύνδεση συμφωνία στο Brexit με μια μεταβατική περίοδο. Προτεραιότητα θα πρέπει να είναι να προστατευτεί το νυν και το επόμενο πι. Για την περίοδο μετά το 2020 όπου είναι αναπόφευκτη η προσαρμογή θα πρέπει να συζητήσουμε όχι μόνο την γεωργική πολιτική μόνη της αλλά να συζητήσουμε ολόκληρο το σύστημα κοινοτικής χρηματοδότησης. Έτσι θα βρεθεί ευκολότερα ένα συμβασμό βέβαιος. Είναι δύσκολη, δύσκολος ο χρονισμός, η στιγμή, η συγκυρία, οπότε πρέπει να αρχίσουμε να τα συζητάμε από τώρα για πράγματα τα οποία έχουν μεγάλη σημασία, π.χ. η ευρωπαϊκή προσταμινή αξία. Και αν γίνει σωστά, είναι μια ευκαιρία να απλοποιηθεί και να βελτιωθεί ο κοινωτικός προϋπολογισμός. Ευχαριστώ. Dobrze, Ευτυχώς που στο τέλος μας είπατε και κάτι θετικό. Αμφίβολης, ε, βέβαια, και αυτό ε, πιθανότητας. Περνάμε στην υποβολή ερωτήσεων. Ο κύριος Άγνιο. Παρακαλώ. σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό που με ανησυχεί με τη μελέτη είναι το τεκμήριο ε, η εικασία ότι οι Βρετανοί φορολογούμενοι, παρόλο που έχουν αποφασίσει να φύγουν, πρέπει να δώσουν ένα τεράστιο ποσό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα πέραν του άρθρου 50 που ήταν ο δικός χάρτης για την έξοδο δεν αναφέρονταν τίποτα για αστρονομικά ποσά που θα πρέπει να δοθούν. Οπότε δεν υπάρχει νομική βάση για αυτό το λογαριασμό του Brexit. Και θα μπορούσα να πω, για να είμαι δίκαιος, ότι θα μπορούσε να ζητηθεί από τους Βρετανούς φορολογουμένους να τιμήσουν τι υποχρεώσει του μέχρι το 2020 και να αναλάβουν τις ευθύνες και για τις συντάξεις των ε, Βρετανών πολιτών που έχουν συνταξιδοτικά δικαιώματα από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το καθεξής. Και τελεία εδώ. Αλλά υπάρχει και μια άλλη όψη στο νόμισμα. Έχουμε ένα σημαντικό κονδύλιο του Βρετανικού στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τι θα γίνει με αυτό. Είχαμε ε, πολλά δάνεια που δώσαμε στις χώρες της Ευρωζώνης, στην Ελλάδα σίγουρα και σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης που είχαν προβλήματα, Πορτογαλία κατά πάσα πιθανόν. Αυτά είναι χρήματα των Βρετανών φορολογουμένων που ήταν, δόθηκαν με τη μορφή δανεισμού, οπότε θα πρέπει να επιστρέψει στη Μεγάλη Βρετανία. Και είμαστε και καθαροί συνεισφορείς. Και έχουμε μετοχικό κεφάλαιο σε ισπανικού αυτοκινητοδρόμου και ιρλανδικέ γέφυρε. Αυτά ήταν χρήματα των Βρετανών φορολογουμένων που χρηματοδότησαν τι υποδομέ και ακόμη βρίσκονται εκεί. Και έχουμε και τις ε, Πρεσβείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά τον κόσμο που έγιναν επίσης με βρετανικά κονδύλια εν μέρη. Επίσης έχουμε τα κτίρια, τα κοινοτικά στο Λουξεμβούργο, Στρασβούργο, Βρυξέλλες. Νομίζω ότι δεν οφείλουμε τίποτα, ούτε ευρώ παραπάνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Κύριε Ευρωβουλευτά. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει ε, να πληρώσει αν ε, δεν τιμήσει υποχρεώσει του το Ηνωμένο Βασίλειο απέναντι σε αυτήν. Ο κύριος Λαζό, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι οι συνέπειες ε, του Brexit στη γαλλική οικονομία. Και μάλιστα σήμερα το εξωτερικό εμπορικό ισοζύγιο τη Γαλλία είναι αρνητικό, με εξαίρεση τα γεωργικά προϊόντα. Σήμερα εξάγουμε προ το Ηνωμένο Βασίλειο 4,5 ε, ε, γεωργικά προϊόντα αξία 4,5 δισεκατομμυρίων. Διόλο μελιτέο ποσό, οπότε ε, μας ενδιαφέρουν οι διαπραγματεύσει με το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί η Γαλλία είναι ζωτική σημασία. Και οι διαπραγματεύσεις αυτές ε, για τον Brexit δεν έχουν ε, ολοκληρωθεί. Δεν έχουμε βρει ακόμη τρόπο για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις εμπορικές συναλλαγές. Θα γίνουν στα πλαίσια της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου, στα πλαίσια μιας τελωνιακής ένωσης ή στα πλαίσια συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών. Αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό, αλλά δεν έχουμε ούτε νομικά ούτε εμπορικά στοιχεία και αυτή η κατάσταση και αυτή η βεβαιότητα είναι ιδιαίτερως ανησυχητική. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ε, υπενθυμίσω και να σας διευκρινίσω ότι οι εμπορικές πτυχές είναι το αντικείμενο της δεύτερης θεματικής ενότητας. Τώρα μιλούμε μόνο για τις δημοσιονομικές πτυχές. Ας επικεντρωθούμε σε αυτό. Ερωτήσεις παρακαλώ και απορίες μόνο για τον προϋπολογισμό, για τις δημοσιονομικές πτυχές. Ο κύριος Φλάνναγκαν. Ευχαριστώ. Προφανώς ως Ιρλανδός ε, Ευρωβουλευτής ενδιαφέρομαι ιδιαίτερο για το θέμα των συνεπειών του Brexit. Άκουσα τα στοιχεία που μας δώσατε και ε, βλέπω πολλά προβλήματα κατά πάσα πιθανότητα. Το θέμα είναι πώς θα τα αντιμετωπίσουμε ε, ήταν ενδιαφέρον το σχόλιο ότι είναι πολιτικό το θέμα. Αν θα γίνουν περικοπές 10 δισεκατομμυρίων, αν θα προέλθουν όλα από τη Γεωργία, θα είναι 3 δισεκατομμύρια το χρηματοδοτικό κενό. Και νομίζω ότι κάτι που θα μα βοηθούσε πολιτικά είναι ε, οι φορολογούμενοι τη Ευρωπαϊκή Ένωση που κατάθεσαν αυτά τα ποσά να νιώσουν ότι έπιασαν τόπο τα χρήματά του. Αν όμω βλέπουν τους βαρώνου του βοηού Κρέατο και το, τη βασιλική οικογένεια ε, να παίρνει χιλιάδες ε, ε, ευρώ σε επιδοτήσεις, τότε δεν θα έχουν αυτή την αίσθηση. Θα πρέπει να ακούσουμε τους φορολογουμένους, τους καταναλωτές. Πώς είναι δυνατόν να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν ένα κοινό γεωργικό προπολογισμό που δεν ευνοεί τους πραγματικούς δικαιούχους, τους παραγωγούς, τους γεωργούς αν θέλουμε να διασφαλίσουμε τον προπολογισμό της κοινή γεωργικής πολιτικής, θα πρέπει να φροντίσουμε να πάει στους ε, γεωργούς, όχι στους μεγάλους κτηματίες ε, ή αυτούς που προσπαθούν να καταστρέψουν τους μικρούς γεωργούς. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να πείσουμε και το λαό και τους ευρωβουλευτέ και το ευρωπαϊκό σύστημα ότι τα κονδύλια που πηγαίνουν στη γεωργία μπορούν να αυξηθούν και όλα ή να μεγιστοποιηθούν. Θα πρέπει όμως να πάνε τα χρήματα αυτά στους πραγματικούς γεωργούς. Αλλιώς δεν θα έχουμε καμία δυνατότητα να προσπίσουμε το γεωργικό προϋπολογισμό. Επίσης, αν μειωθεί ο προϋπολογισμός του ΣΚΑΠ, θα πρέπει τα κονδύλια που θα απομείνουν να πάνε στους μικρούς καλλιεργητές, στους μικρούς γεωργούς, στους πραγματικούς γεωργούς, αυθεντικούς. Έχουμε μια κατάσταση που επαναλαμβάνεται από πολλές ομάδες. Φαίνεται ότι όλοι το δηλώνουν. 80% των κονδυλίων της ΚΑΠ πηγαίνει στο 20% των γεωργών. Αν γίνουν ε, περικοπές, οι περικοπές να γίνουν σε αυτούς που παίρνουν το 80% των κονδυλίων και να αφήσουμε αυτούς που καρπώνονται μόνο το 20% του πραγματικού γεωργού ε, το ποσό του άθικτο. Οπότε μόνο αν πηγαίνουν στους πραγματικούς γεωργούς δεν θα πηγαίνουν στους ε, κερδοσκόπους αυτά και αυτό θα είναι το καλύτερο. Κύριε Φλάνακαν θα σας παρακαλούσα να μην κάνετε σχόλια εκτός θέματος. Και το πού πηγαίνουν τα κονδύλια της ΚΑΠ δεν είναι αντικείμενο της σημερινής συζήτησης. Αυτό το συζητήσουμε αλλού. Εδώ μιλούμε για τις δημοσιονομικές πτυχές ε, και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις του Brexit. Παρακαλώ να εστιαστούμε στο θέμα της σημερινής συζήτησης. Ο κύριος Ντες. Ο κύριος Ντες. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ τους δύο ομιλητές μας για τις παρουσιάσεις. Είναι ξεκάθαρο ότι τώρα που το Ηνωμένο Βασίλειο θα υπάρχουν λιγότερα χρήματα. Αυτό είναι σαφές. Το τι συνέπειες θα φέρει στην γεωργική πολιτική μπορούν να το αναλύσουν διαφορετικά σενάρια. Αλλά ένα πράγμα δεν μπορεί να συμβεί ότι η μείωση των εσόδων δεν θα πρέπει να είναι εις βάρος του τομέα της γεωργίας μόνο. Όποια μείωση σε έσοδα, σε ποσά διαθέσιμα θα πρέπει αναλογικά να επιβαρύνει κάθε τομέα του προϋπολογισμού. Αυτό είναι το πρώτο μου πολιτικό μήνυμα. Τώρα μετά πώς θα γίνει η κατανομή των ποσών συγκεκριμένα είναι μια άλλη συζήτηση και δεν έχω αρκετό χρόνο για να την αναπτύξω. Αλλά για τους δύο μιλητές μας έχω την εξή ερώτηση. Βλέπετε μια δυνατότητα, και πάλι είναι πολιτικό βέβαια το ερώτημα, να εξασφαλιστούν από κάπου επιπλέον χρήματα, γιατί δεν γίνεται βέβαια τα κράτη-μέλη να προσφέρουν περισσότερα ποσά ε, να αναθέτουν περισσότερες δαπάνες, περισσότερα ε, καθήκοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς όμως να αυξάνουν και τη συνεισφορά τους. Και νομίζω ότι θα πρέπει να μεριμνούμε έτσι ώστε όταν αναλαμβάνει περισσότερα καθήκοντα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα της προσφέρεται και κατάλληλη χρηματοδότηση. Ο Υπουργό των Οικονομικών Σόιμπλε, για πολλά χρόνια Υπουργό των Οικονομικών, έκανε σαφεί δηλώσει πριν από μερικού μήνε εδώ γιατί είτε πρόκειται για την προστασία των εξωτερικών συνόρων, είτε πρόκειται για άλλους τομείς η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να εξασφαλίσει και κατάλληλη πρικοδότηση. Εμείς εδώ στην Επιτροπή Γεωργίας δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε αυτά τα προβλήματα, είναι θέματα του προϋπολογισμού, των συναδελφών της Επιτροπής των Προϋπολογισμών και βέβαια των κρατών μελών. Εσείς μας επισημαίνετε τι είδους συνέπειες μπορεί να προκύψουν από αυτή την αλλαγή για τον κύριο Άγνιου. Θέλω να πω πως ιδιαίτερα φοβούμε πως θα προκύψουν από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου σημαντικές τρευλώσεις του ανταγωνισμού σε σχέση με τα γεωργικά προϊόντα. Γιατί, μέχρι, γιατί από ό,τι φαίνεται οι γεωργοί του Ηνωμένου Βασιλείου θα παίρνουν διπλές επιστροφές από ό,τι μέχρι τώρα. Και προφανώς θα υπάρχουν σοβαρές τρευλώσεις του ανταγωνισμού. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστώ τους δύο προσκεκλημένους για τις τοποθετήσεις τους για τον ε, προϋπολογισμό και συμφωνώ εδώ με τον Αλμπερτές. Αναφέρεσαι σε τρία διαφορετικά σενάρια. Είτε αυξάνουν τις συνεισφορές, τα κράτη-μέλη, είτε μειώνονται οι δαπάνες, είτε συνδυάζονται τα δύο. Αλλά, αν κατάλαβα καλά, αλλά για ιδίους πόρους δεν μας λέτε τίποτα. Και όμως ένα πραγματικό ζήτημα στο οποίο θέλω ακριβώς να σας διατυπώσω το ερώτημα. Γιατί το επιλέξατε. Ή το έχετε αφήσει κατά μέρος το θέμα αυτό και το αγνοείτε. Τώρα είμαστε στο φαινόμενο της ψαλίδας, ότι δηλαδή δεν μπορούμε να αποκόψουμε το Brexit, την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, από την περικοπή των εσόδων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν οι μεγάλες πολιτικές, τα θέματα της άμυνας, της αντιμετώπισης της ε, μετανάστευσης, ε, της ε, κοινωνικής και φορολογικής εναρμόνισης. Άρα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το φαινόμενο αυτό της ψαλίδας που θα μας θέσει ενώπιον το αμήλικο του ερωτήματος τι δομές θέλουμε, τι θέλουμε εμείς αν δεν αυξήσουμε την ε, συνεισφορά των κρατών μελών με τον κανόνα του 1% και δεν δώσουμε ιδίους πόρους, δεν θα είναι σε θέση να επιτελέσει το έργο της να εκτελέσει τα καθήκοντά της Ευρωπαϊκή Ένωση. Είτε πρόκειται για περικοπές στην συνοχή ή για, τη, για περικοπές στην ΚΑΠ, πάλι δεν πρόκειται να δώσουμε καμιά απάντηση ουσιαστική. Και ναι, είναι πολύ συγκεκριμένα γεωργικό το πρόβλημα συνέπειας, δηλαδή για τη γεωργία θα υπάρξουν οπωσδήποτε, αλλά όχι μόνο, είναι πολύ γενικότερο ταυτόχρονα. Αυτό ήθελα να επισημάνω για να διευρύνετε λίγο τον ορίζοντα το, της θεματολογίας σας. Στη μεταρρύθμιση τώρα της ΚΑΠ μας λέτε ότι δεν υπάρχει τεχνική μέθοδος για την προσμέτρηση των συνεπειών του Brexit στο μέλλον, στη μελλοντική μεταρρύθμιση. Δηλαδή μας λέτε ότι δεν πρέπει να σκεφτούμε το δημοσιονομικό πρόβλημα, στο οποίο δεν δίνονται μακροπρόθεσμα απαντήσεις, και μας καλείτε να, κάνουμε, να επεξεργαστούμε το θέμα μόνο μέσα από ένα πολιτικό όραμα. Μα νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για την ουσία. Όταν άλλες ήπειροι και δυνάμεις όλο τον κόσμο αυξάνουν τους προϋπολογισμούς για την πολιτική, τη γεωργική ή των τροφίμων, δεν είναι δυνατόν να υπολείπεται ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός των αναγκών ακόμη. Πρέπει να μιλήσουμε βεβαίω για τα τεχνικά ζητήματα, αλλά δεν είμαστε εδώ, δεν μπορούμε να κάνουμε μόνο μηχανιστικές, ε, ε, να δίνουμε μόνο μηχανιστικές λύσεις, πρέπει να μιλήσουμε για την ουσία. Και πρέπει και η Επιτροπή να αναλάβει να συζητήσει το έργο, το πρόγραμμα, το σχεδιασμό μιας μελλοντικής γεωργικής πολιτικής. Παρακαλώ, όχι πάνω από δύο λεπτά ο καθένας. Βλέπετε το χρονόμετρο μπροστά σα. Δέκα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του χρόνου θα σηκώνω το ε, σφυράκι μου. Κυρία Αγγιλέρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ερχόμαστε στα συγκεκριμένα γιατί ε, και ο κύριος Δες και ο κύριος Αντριέ με πρόλαβα. Ποια είναι η γνώμη σας, γιατί δεν μας είπατε από ό,τι βλέπω, τι γίνεται με την απώλεια των χρηματο... χρηματοδοτήσεων. Μας είπατε ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι συνεισφορές ή να γίνουν περικοπές ή να μην έχουμε συμφωνία. Εμείς όμως ως ομάδα εξετάζουμε και την πιθανότητα ιδίων πόρων. Δηλαδή να αυξηθούν ήδη ίδιοι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κάποιους ε, ειδικού κοινοτικού φόρους που θα αυξάνουν τα κοινοτικά κονδύλια και θα τροφοδοτούν τον ευρωπαϊκό, τον ενωσιακό προϋπολογισμό. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτή την πτυχή που δεν την ε, α, αναφέρατε. Δεν ξέρω αν τη λάβατε υπόψη. Δεν θα μπορούσαμε με αύξηση των ιδίων πόρων, με τη θέσπιση ενό ειδικού φόρου, να καλύψουμε ένα τμήμα του χρηματοδοτικού κενού. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Επίσης, ε, μας είπατε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει και τις ε, πληρωμές του Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων για το 2019 και 2020. Αυτό με θορύβησε, εκτός αν δεν σας άκουσα καλά. Δεν είπατε για, για το Γεωργικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, αλλά για τις εγγύησεις, ε, τις πληρωμές του πρώτου πυλώνα, δηλαδή τις άμεσες ενισχύσεις. Κάτι τέτοιο, αν το έβλεπαν στις εφημερίδες, θα, θα τρομοκρατούσε τους ε, παραγωγούς δηλαδή να επηρεαστούν οι πληρωμές των άμεσων ενισχύσεων για το 2019 ή 2020 λόγω Brexit. Θα πρέπει να το εξηγήσουμε καλά για να μην δημιουργήσουμε αβεβαιότητα και πανικοβάλλουμε τους ε, γεωργού. Παρακαλώ. Θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι κάποιες ερωτήσεις ε, είναι περισσότερο για πολιτικούς ηθήνοντες, όχι για εμπειρογνώμονες. Οπότε καλό θα κάνουμε ένα διαχωρισμό. Η κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους ειδικού για τα νούμερα. Όλα τα ζητήματα είναι πολιτικά και δεν μπορούν να τα απαντήσουν οι εμπειρογνώμονες, αλλά έχω να κάνω μια παρατήρηση για τη διαφάνεια που έλεγε για τις επιδράσεις που θα υπάρχουν άπαξ που λέτε ότι δεν θα πρέπει να συνδέσουμε το Brexit με κάποιες υποθετικές μεταβατικές διατάξεις. Έχετε μείνει πίσω όμως γιατί από ό,τι ακούω από τους διαπραγματευτές ε, ιδιωτικό και δημοσίω. Αυτή τη στιγμή το Ηνωμένο Βασίλειο συνδέει την πληρωμή των δεσμεύσεών του με την τελική συμφωνία, οπότε έχουν προχωρήσει παρακάτω. Με ενδιαφέρον άκουσα και τον συνάδελφο τον κύριο Άγνιο. Ε, και ας κανχάζει γιατί πραγματικά μας δίνει την αίσθηση του τι αντιμετωπίζουμε. Και σέβομαι βεβαίως ε, τα όσα ξέρει για τη γεωργία, αλλά όχι τόσο αυτά τα οποία έχετε ως αλληλεγγύη. Και τα σχόλιά σας εδώ, και βεβαίως υπάρχει ελευθερία λόγου, ε, δείχνουν μια περιφρόνηση για την έννοια της αλληλεγγύης. Και όταν μιλάτε για τις γέφυρες στην Ιρλανδία, πραγματικά, ε, πολύ κακό γουστό. Ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρώπη ακριβώ έχει ω αντικείμενο την αλληλεγγύη μεταξύ λαών, έτσι ώστε αυτοί οι οποίοι έχουν λιγότερα να μπορούν να αναπτυχθούν και να γίνουν ισχυρότεροι. Αυτό είναι η Ευρώπη. Αν δεν το έχετε καταλάβει, ίσω γι' αυτό θέλετε να φύγετε. Αλλά να μα μεταχειρίζεστε με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Ο κ. Νίκολσον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πρόκληση είναι τεράστια, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να δούμε την πραγματικότητα. Όταν ο κύριος Μπαρνιέ μίλησε ενώπιον του Ιρλανδικού Κοινοβουλίου και στην Ιρλανδία έχουμε μάλλον τη δυσκολότερη κατάσταση γιατί τα σύνορα αυτή τη στιγμή εκεί είναι μεταξύ της Βορείου Ιρλανδίας και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας αλλά όταν θα φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνουν τα σύνορα μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, είναι άρα μεγάλη η διαφορά και ο κύριος Μπαγκίνη ότι θα υπάρξουν συνέπειες, προβλήματα. Ε, δυσκολίες. Για ε, τον κύριο Άγνιου θα το έλεγα το εξής. Ε, σπανίως συμφωνώ με την πρόεδρο του κόμματο τους. Αλλά πριν από λίγους μήνες έβγαλε μια ομιλία στο Στρασβούργο ο πρόεδρος σας και είπε τότε στον κύριο Γιούνκερ εάν είχατε δώσει κάτι στον πρόεδρο Κάμερον για να παλέψει το δημοψήφισμα, δεν θα ήταν αυτό το αποτέλεσμα. Και οφείλω να πω ότι συμφωνώ με αυτό. Εδώ βρισκόμαστε σήμερα λόγω της αδιαλαξίας του παρελθόντος. Οπότε ας μην επιτρέψουμε στην αδιαλαξία του παρελθόντος να υπαγορεύσει το μέλλον. αν υπάρξει πρόβλημα με το Ρωμανό στην έξοδο θα ε, έχουμε καταστροφή για όλα τα μέρη. Άκουσα με ενδιαφέρον όσα είπαν οι ειδικοί εδώ. Αλλά η κυρία... Ε, δυστυχώς δεν με βοηθάνε τα μάτια μου να δω το όνομά σας. Ανέφερε κάτι και θα ήθελα να μας το εξηγήσει η μίληση για αλλαγή στη δυναμική των διαπραγματεύσεων. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ε, ακριβώ ε, σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι η εξουσία από τις βόρειες χώρες θα πάει στις νότιες χώρες της Ευρώπης. Και τι ε, σημαίνει αυτό και προς τον κύριο Χάς είπε για τον προπολογισμό. Ότι εάν το χειριστούμε σωστά μπορεί να απλοποιηθεί ο κοινοτικό προπολογισμό. Μπορείτε να μα το εξηγήσετε αυτό. Πώ θα γίνει αυτό, γιατί εγώ δεν θέλω όταν θα φύγουμε εμεί ω Ηνωμένο Βασίλειο, δεν θέλω να διαλυθεί α, ε, η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριο Σκάρθη. Thank you, um, Chair. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Χαίρομαι που γίνεται αυτή η συζήτηση με το Policy Department και την έκθεσή τους, διότι βλέπω ότι ως Επιτροπή σε πολλά θέματα ε, υστερούμε, ερχόμαστε με καθυστέρηση να αντιμετωπίσουμε τις ε, δονήσεις που προξενεί το Brexit, το κλον, τους κλονισμούς καλύτερα. Και βέβαια η κατάσταση θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο, αυτό το έχουμε δει και στην Ιρλανδία. Είναι ασφαλώς ζωφερή η εικόνα του μέλλοντος για το γεωργικό τομέα. Για την Ιρλανδία συγκεκριμένα είναι σαφές ότι θα έχουμε σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις. Εάν δούμε τους ε, τομείς πολιτικής και στα 28 κράτη-μέλη βλέπουμε ότι αυτοί που θα αυτοί που, έχουν υποστεί, που θα υποστούν τις σοβαρότερες συνέπειες θα είναι γεωργοί και για το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και για την Ιρλανδία όπως και για όλες τις άλλες χώρες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Το Κοινοβούλιο έχει υιοθετήσει σαφείς θέσεις για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες του Brexit και πρέπει η Επιτροπή μας να δείξει σκληρή στάση, δεδομένου ότι απειλείται από μια καταστροφή ο γεωργικός τομέας και δεν νομίζω ότι υπερβάλλω, γιατί και τα κοινά σύνορα και η γεωγραφική ε, εγκύτητα, αλλά και η φύση της ε, Ιρλανδίας ως νησιού οδηγεί σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα γεωργίας και άρα οι συνέπειες από την καταστροφή αγορών, από την απώλεια αγορών, είτε στο βορρά είτε στο νότο του νησιού, θα φέρουν και στην άλλη πλευρά καταστροφικές συνέπειες. Κάθε ή μάλλον μεγάλο ποσοστό των γεωργικών εξαγωγών της Ιρλανδίας περνάει μέσα από την ίσο της Βρετανίας και αυτό θα έχει σοβαρές συνέπειες. Πάνω απ' όλα λοιπόν πρέπει να είμαστε ενήμεροι για τους κινδύνους και πρέπει να ορίσουμε τις θέσεις του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με την Βόρεια Ιρλανδία. Και βέβαια πρέπει να, πρέπει να προστατέψουμε την ίσο της Ιρλανδίας γιατί οι συνέπειες θα είναι τεράστιες. Ευχαριστώ κύριος Μπράνεν. Ευχαριστώ. Ως κάποιος από τους Βρετανούς που τάχθηκαν υπέρ του, της παραμονής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, βλέποντας τη, τα ομά νούμερα της μελέτης, Πραγματικά λυπάμαι ακόμη περισσότερο που χάσαμε το δημοψήφισμα γιατί βλέπω, βλέπω τις επιπτώσεις ε, και τους αριθμούς που μιλούν από μόνο τους. Ε, βλέπω τη γυμνή πραγματικότητα και λυπάμαι γιατί πραγματικά ε, οι συνέπειες θα αγγίξουν το απλού πολίτε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Μαρέτ μίλησε για την αλληλεγγύη, πολύ σωστά, γιατί η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου υπονομεύει αυτή την ε, αλληλεγγύη γιατί θα μείνουν λιγότερα κονδύλια στον ενωσιακό προπολογισμό. Και θα ήθελα να ζητήσω και ένα συγγνώμη από τη Δημοκρατία τη Ιρλανδίας, γιατί θυμάμαι όταν πήγαινα μικρό παιδί να ψωνίσω με τη μαμά μου, μου έλεγε ότι χρειαζόμασταν βούτυρο και πήγαινα στο ψυγείο να, να πάρω βούτυρο και μου λέει όχι αυτό το βούτυρο, το Ιρλανδικό βούτυρο εγώ πάρε και τη ρωτούσα γιατί αγοράζουμε μαμά Ιρλανδικό βούτυρο και μου είπε μετά από αυτά που έχουμε κάνει εμείς οι Άγγλοι στους Ιρλανδούς το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αγοράζουμε το βούτυρό τους και αυτό πραγματικά ήταν ένα μάθημα ιστορίας που έμαθα τότε και επίσης έχω μία ερώτηση ε, ε, τα νούμερα που μας δώσετε για την επίπτωση στις επιμέρους χώρες Ας μην ξεχνούμε ότι αφορούν την παραγωγή τροφίμων. Έχετε ασχοληθεί καθόλου ή γνωρίζετε κάποιες μελέτες που αφορούν την ε, παραγωγή τροφίμων, αν μειωθεί κατά 10% η παραγωγή, σημαίνει ότι θα παράγουμε κατά 10% λιγότερα τρόφιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν ξοδεύουμε λιγότερα κονδύλια στην κοινή γεωρική πολιτική, δεν θα οδηγηθούμε μοιραία στον περιορισμό της παραγωγής τροφίμων. Και δεν θα πρέπει να πούμε και στο κοινό τι θα συμβεί, γιατί ε, θα πρέπει να δώσουμε ένα ποσοστό. Τι θα σημαίνει ε, ένα τέτοιο ποσοστό στον περιορισμό της παραγωγής τροφίμων. Θα είναι μια χρήσιμη πληροφορία που χρειαζόμαστε εμείς οι Ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ κύριο Μπόγκοβιτς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για τις μελέτες που μας παρουσιάσατε. Είναι πολύ χρήσιμα αυτά τα στοιχεία που μας έδωσαν οι εμπειρογνώμονες. Εγώ Φυσικά είμαι πάντα υπέρ της ανάλυσης των συνεπειών των πράξεών μας. Δυστυχώς, κάπως καθυστερημένα μας έρχονται αυτές οι μελέτες. Θα έπρεπε να τις είχαμε λάβει πριν να ληφθούν κάποια μέτρα για τον Brexit. Εν πάση περιπτώσει είναι σίγουρο ότι θα έχουμε επιπτώσεις και δημοσιονομικές και εμπορικές σε ό,τι αφορά την ροή των εμπορικών συναλλαγών. Εμείς ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εντείνουμε τις συζητήσεις για τον Brexit. Έχουμε τις διαπραγματεύσεις, έχουμε το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τη διαμόρφωση της μελλοντική κοινή γεωργικής πολιτικής. Αναφυσβήτητα όλες αυτές οι πολιτικές και όλες αυτές οι συζητήσεις επιδέχονται βελτιώσεις και το Brexit θα μας δώσει ευκαιρία για να προβληματιστούμε για τη χρησιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τι στηρίζεται αυτή. Στηρίζεται στην αλληλεγγύη. Στην αλληλεγγύη με τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και δεν θα πρέπει επίσης να ξεχνούμε ότι όταν έχουμε μία ελεύθερη αγορά εποφελούνται και οι καθαροί εξαγωγείς. Ελπίζω όλα αυτά τα στοιχεία να ληφθούν υπόψη στη συζήτηση και να πρετανεύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση η αρχή της αλληλεγγύης. Πιστεύω ότι όλα όσα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν περιορίζονται σε αυτό το 1%. Ίσως θα έπρεπε να επιτύχουμε το 1,23% που επιτρέπει η συνθήκη της Λισαβόνας. Θέλουμε μια αλληλέγγυα με τους πολίτες Ευρωπαϊκή Ένωση για να θέλουν οι πολίτες να παραμείνουν σε αυτήν. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Θα ξαναδώσω το λόγο στους εμπειρογνωμονές μας, στους καλεσμένους μας, για να απαντήσουν στις ερωτήσεις. Ε, οι δυο μαζί 10 λεπτά, αλλά όχι παραπάνω παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις σας και νομίζω ότι μπορώ να απαντήσω μερικές από αυτές ομαδοποιημένες, καθώς κάποιοι από σας αναφερθήκατε στην δυνατότητα για εξασφάλιση νέων πόρων από είτε ιδίου πόρους είτε άλλες συνεισφορές. Αλλά, πολύ σύντομα, ας απαντήσουμε στο ερώτημα το σχετικό με την ε, παραγωγή τροφίμων. Ο καθηγητή Μάθιου είναι πολύ πιο ειδικό από μένα και θα σα δώσει μια αξιολόγηση, μια εκτίμηση μάλλον, στην βελτίωση των δαπανών. Βεβαίω και θα βοηθήσει αυτό. Στην ε, βελτίωση της ανοχής για υψηλότερες δαπάνες ε, στα νέα κράτη και κυρίως στα κράτη που συνεισφέρουν καθαρά στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Αλλά ίσως θα έπρεπε να γίνει μια μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων και αναφέρεται στις συστάσεις μας. Ο Μάριο Μόντι και η ομάδα εμπειρογνωμόνων δημοσίευσαν σε αρχές του χρόνου ε, μια έκθεση για τη μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων ε, και την αναδιαμόρφωσή του έτσι ώστε να λάβει υπόψη τις συνέπειες του Brexit. Δυστυχώς όμως δεν ε, έτυχε της προσοχής που θα άξιζε αυτή η έκθεση. Υπάρχει λοιπόν δουλειά περαιτέρω, αλλά ταυτόχρονα πρέπει και να διευκρινιστεί ότι οι εθνικές συνεισφορές συνιστούν ιδίους πόρους. Με την εισαγωγή νέων ιδιών πόρων, δεν αλλάζει το σύστημα των καθαρών υπολείπων ή μη. Δηλαδή και με μια μεταρρύθμιση του σύστηματος των ιδιοπόρων, απλώς θα μειωθούν αντίστοιχα οι συνεισφορές των κρατών μέλων. Δεν θα έχει περισσότερα χρήματα προπολογισμό. Και βέβαια η έκθεση Μόντι είχε πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες γιατί μιλούσε για ένα φόρο του διοξιδίου του άνθρακα, ένα φόρο του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά μην ξεχνάτε ότι κάθε φορά τα κράτη-μέλη θα το χαρακτηρίζουν ίδιο πόρο και θα το αφαιρούν από, τις, ε, από τα ε, ποσά που συνεισφέρουν, από τα καθαρά υπόλοιπα μόνο αν δεχθούν ότι είναι συμφέρον ολόκληρης Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δεχθούν την αύξηση των εισφορών τους. Και τελευταίο, από την διαφάνεια της σχετική με την αύξηση των συνεισφορών. Βλέπουμε ότι δεν θα είναι τεράστιες ε, οι αυξήσεις των συνεισφορών των κρατών μελών, αλλά πολιτικά θα έχουν μεγάλο ειδικό βάρος, θα επηρεάσουν σημαντικά την πολιτική ζωή των κρατών μελών και ιδιαίτερα των καθαρών συνεισφορέων. Και το έχουμε ήδη δει από τη Γερμανία, από την Αυστρία. Οι πρώτες αντιδράσεις ήταν ε, εξ αρχής, δεν πρόκειται να δώσουμε παραπάνω από όσα ήδη συνεισφέρουμε. Ε, ίσως θα ήταν αυτό μια ευκαιρία για απλοποίηση του συστήματος του δημοσιονομικού, γιατί θα μπορούσαν έτσι αφού τελειώνει μια επιστροφή να τελειώσουν όλες, πράγμα το οποίο θα ήταν καλό. Από την άλλη είναι δύσκολο ταυτόχρονα με την, με την αύξηση των συνεισφορών να επιβληθεί η κατάργηση των επιστροφών, διότι και θα πληρώνουν περισσότερα οι καθαροί συνεισφορείς και θα τους αφαιρεθεί η έκπτωση, η επιστροφή. Αυτό θα είναι δύσκολο να περάσει δηλαδή. Για το θέμα των ιδίων πόρων συνεχίζω. Το αναφέρουμε και στη μελέτη μας και σίγουρα πολλές προσδοκίες υπάρχει για αυτό το σενάριο, την πιθανότητα αύξηση των ιδιών πόρων. Και φυσικά στην πρόταση μας και το Ίδρυμά μας, Ζακ ε, Δελόρ, είναι υπέρ και είχαμε πολλά έγγραφα στα οποία ζητούσαμε μεταρρύθμιση του συστήματος ιδιών πόρων, γιατί αυτό θα είναι ε, το καλύτερο για το μέλλον της Ευρώπης, να μεταρρυθμίσει το σύστημα, το σύστημα ιδιών πόρων της ε, αλλά δεν ξέρω αν είναι δυνατή κάποια ρηξικέλευθη τέτοια μεταρρύθμιση για τους ιδίους σπόρους πριν το 2020. Και αν δείτε το έγγραφο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού, έχω την αίσθηση ότι ε, θεωρεί ότι η δημιουργία νέων πόρων είναι ο εύκολος τρόπος για να μετριαστούν οι συνέπειε του Brexit πάντα αναφέρονται το θέμα των μεταρρυθμίσεων των ίδιων πόρων, αλλά αν δείτε πόσο χρόνο χρειάστηκε για να κυρωθεί το θέμα των ίδιων πόρων, ήταν τρία χρόνια. Ε, το 2009, 2011 ε, μάλλον ε, υποβλήθηκε, το 2014 εγκρίθηκε. Τώρα έχουμε μόνο 1,5 χρόνο για να διαπραγματευτούμε και να κυρώσουμε ένα νέο σύστημα ιδίων πόρων και το προηγούμενο δεν δημιούργησε πολλές μεγάλες αλλαγές. Δεν περιληφθήκε πραγματικά νέος ίδιος πόρος, οπότε είμαι κάπως απεσιόδοξο προς την ικανότητα να θεσπίσουμε νέο ίδιο πόρο που πραγματικά θα τροφοδοτήσει το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και μάλιστα τόσο γρήγορα μέχρι το 2020, τόσο σύντομο χρόνο χρονικό διάστημα. Μπορεί να υλοποιηθεί αυτό το σενάριο, αλλά όχι τόσο σύντομα, όχι μέχρι το 2020. Οπότε θα σας πρότεινα ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ετοιμαστείτε, να μην ε, είναι έτοιμος αυτός ο νέος εύκολος, πιο Τρόπο προσαρμογή μέχρι το 2020. Οπότε θα χρειαστεί να κινητοποιηθούν τα πιο δύσκολα σενάρια, δηλαδή η αύξηση των συνεισφορών, η μείωση των δαπανών, που μπορεί να είναι πιο δυσεφάρμοστα, αλλά είναι πιο ρεαλιστικά. Δεν είναι ότι είμαστε κατά των ιδίων πόρων, αλλά για να είμαστε ρεαλιστέ από πολιτική άποψη, δύσκολο είναι σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να γίνει διαπραγμάτευση και να ε, προταθεί ένα νέο σύστημα ιδίων πόρων. Αν θυμάστε το τελευταίο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και όλες τις τελευταίες διαπραγματεύσεις, το Ηνωμένο Βασίλειο ενέκαθεν ήταν ε, η χώρα με την πιο ακραία θέση ε, που ήταν στην ομάδα των καθαρών συνεισφορέων. Είχε την πιο ριζοσπαστική προσέγγιση και στις τελευταίες διαπραγματεύσεις εξαιτίας του Ηνωμένου Βασιλείου είχαμε τόσο χαμηλό συνολικό ανατοτόριο πληρωμών. Για τελευταία στιγμή το Ηνωμένο Βασίλειο ζήτησε να μειωθεί το επίπεδο πληρωμών του ΠΔΠ. Και αυτό είναι ηρωνικό να το σκεφτείτε. Γιατί αν έχουμε μεγάλο ράλκα ε, η προς εκαθάριση ε, στο ΠΔΕΛΤΑΠ είναι ε, χάρη στο Ηνωμένο Βασίλειο που μείωσε αισθητά το επίπεδο πληρωμών του, του ισχύοντος πι. Οπότε το Brexit ε, ίσως αλλάξει τη δυναμική των διαπραγματεύσεων μεταξύ των καθαρών συνεισφορέων. Δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Ίσως έχουμε μια πιο επικοδομητική προσέγγιση, ακόμη αν θα είναι πιο δύσκολο, γιατί με το χρηματοδοτικό καιρό του Brexit ίσως υποβληθούν ε, απαιτήσει για αύξηση των συνεισφορών. Θα δούμε. Πάντω αλλάξει η δυναμική των διαπραγματεύσεων σίγουρα. Σε ό,τι αφορά τη συμφωνία για το Brexit, ίσω το πιο εύκολο είναι αυτά τα δύο γεωρικά ταμεία τη αγροτική ανάπτυξη και των εγγύσεων και πώ θα επηρεαστούν. Στι αρχικέ διαπραγματεύσει για τον Brexit είχαμε δύο θέσει ω προ το πώ ε, οι δαπάνε και η αναλήψη υποχρεώσεων ε, που περιλαμβάνονται στο ΠΔΕΛΤΑΠ αλλά δεν έχουν εγγραφεί στου αιτήσου προπολογισμού, αν θα περιλαμβάνονται στο λογαριασμό του Brexit. Μερικοί είπαν μόνο οι δεσμεύσει ε, δαπανών που δεν έχουν εγγραφεί στου αιτήσου προπολογισμού ε, να περιληφθούν. Και αυτέ που είναι στου ενοποιημένου λογαριασμού και θεωρούνται υποχρεώσει. Δηλαδή αυτέ που ήδη έχουν μεταφραστεί σε συμβάσει. Αυτέ οι υποχρεώσει που για τις οποίες υπάρχουν ε, ε, συμβάσεις. Δηλαδή έχουμε την Επιτροπή και έναν ε, δικαιούχο. Συνήθως είναι τα διαρθρωτικά ταμεία με προγράμματα και συγκεκριμένους δικαιούχους. Και στους ενοποιημένους λογαριασμούς ήδη αυτά θεωρούνται υποχρεώσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα αυτό είναι ίσονος σημασία, γιατί οι πληρωμές ΚΑΠ δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις υποχρεώσεις πληρωμών και είναι ίσονος σημασία γιατί μετά την ομιλία της Θερέζα Μέη που αποδέχτηκε, συμφώνησε ε, ή τουλάχιστον ανέλαβε τη δέσμευση να καλύψει όλες τις καθαρές συνεισφορές ε, του Ηνωμένου Βασιλείου μέχρι το τέλος του ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ, οπότε το θέμα δεν θα είναι σημαντικό. Το θέμα είναι κατά πόσο το Ηνωμένο Βασίλειο θα συμμετέχει και στις πληρωμές των ε, εκκρεμών υπολείπων προς εκαθάριση του 2020. Επίση, αναφέρθηκαν οι νομικέ πτυχέ, οι νομικέ υποχρεώσει του Ηνωμένου Βασιλείου να καταβάλει το λογαριασμό του Brexit. Ε, το Ηνωμένο Βασίλειο φαίνεται δεν κατάλαβε τη φύση αυτού του λογαριασμού, γιατί από την αρχή η θέση του ε, Ηνωμένου Βασιλείου ήταν ε, αμυγός νομικίστικη, αλλά δεν είναι τόσο νομική η πτυχή του λογαριασμού του Brexit, είναι περισσότερο πολιτική. Και ουσιαστικά ε, το Ηνωμένο Βασίλειο ζητήθηκε να συμμετέχει για να γίνει με έφτακτο τρόπο αυτή η αποχώρηση και να μην δυσχεράνει την κατάσταση των υπόλοιπων κρατών μελών. Γιατί θα δημιουργηθεί μεγάλο χρηματοδοτικό κενό λόγω Brexit και μετά το ΠΔΠ. Οπότε είναι λογικό και είναι θέμα πολιτικής ευθύνης για το Ηνωμένο Βασίλειο, για το κράτος μέλος που αποχωρεί, να μην κάνει τη ζωή πολύ δύσκολη, ε, τουλάχιστον για τον ΙΝ ΠΔΠ, για τους υπόλοιπους. Τώρα αρχίζει κάπως ε, να αναγνωρίζεται αυτή η υποχρέωση μετά την ομιλία της Φλωρεντίας της Θερέζα Μέη. Κατάλαβε δηλαδή ότι δεν είναι τόσο νομική αλλά πιο πολιτική προσέγγιση. Δεν θέλουμε εξαιτία μα να δυσκολευτούν όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Αλλά ε, το συνδέει ω προπόθεση με τη μεταβατική συμφωνία το θέμα του λογαριασμού. Και σίγουρα αυτή η διασύνδεση είναι κάτι που ζητά το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά δεν έχει γίνει ακόμη δεκτό. Δηλαδή το να συνδέσουμε το λογαριασμό του Brexit με τη μεταβατική συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμη δεν το δέχεται. Και η προσωπική μου άποψη είναι ότι υπάρχει κάποιο είδος άδεια που δίνουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο να συνδέσει για την Βρετανική κοινή γνώμη το λογαριασμό με τη μεταβατική συμφωνία, αλλά δεν νομίζω ότι στην πορεία θα, συνδεθούν, θα συνδεθεί το θέμα του λογαριασμού με τι οποιοδήποτε μεταβατικέ συμφωνίε. Κάτι που θα είναι πολύ αρνητικό αν γίνει αυτή η σύνδεση για την, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τη γνώμη μου. Σας ευχαριστώ. Και περνάμε στο δεύτερο σκέλος, στη δεύτερη θεματική ενότητα τις εμπορικές πτυχές, γεωργικές συναλλαγές Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου. Ε, θα έχουμε ως ομιλητές την κυρία Σεσίλια Μπελόρα και τον κύριο Ζαν Φουγέ από το Κέντρο Διεθνούς ε, Έρευνας και Οικονομικού Σχεδιασμού του Παρισιού. 20 λεπτά έχετε κι εσείς. Θα επικεντρωθούμε στις εμπορικές πτυχές, στο γεωρικό εμπόριο Ευρωπαϊκής Ένωση Ηνωμένου Βασιλείου και παρακαλώ στις γεωρικές πτυχές και στο γεωρικό εμπόριο να περιοριστούν και οι ερωτήσεις των συναδέλφων. Έχετε 20 λεπτά παρακαλώ, οι δύο εμπειρογνώμονέ μας για το δεύτερο σκέλος. Παρακαλώ ξεκινήστε. Καλημέρα και ευχαριστώ για την προσοχή σας. Θα παρουσιάσω τα κύρια ευρήματα της έκθεσης. Ανάλυση των τρέχουσων εμπορικών σχέσεων μεταξύ των 27 και του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο συνάδελφος Αμφουγάς στη συνέχεια θα σας παρουσιάσει μια επισκόπηση των κύριων ε, συνεπειών μετά το Brexit, εάν δεν υπάρχει συμφωνία με τον Ηνωμένο Βασίλειο. Οι στατιστικές λοιπόν, οι εμπορικές, ε, μπορούν να μας δώσουν πολλές πληροφορίες για το ποιες θα μπορούσαν να ήταν οι χώρες ή οι τομείς που θα επηρεαστούν περισσότερο από το Brexit. Αν κοιτάξουμε τα στοιχεία, συγκεκριμένα το πρώτο σημείο, που, το πρώτο χαρακτηριστικό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει απουσία συμμετρίας Ε, είναι μια χώρα με, σημαντικό, με σημαντικά νούμερα και σε ΑΕΠ και σε πληθυσμό βέβαια το Ηνωμένο Βασίλειο τρίτο σε πληθυσμό, άρα αντιλαμβανόμαστε τι είδου αγορά ε, αντιπροσωπεύει. Αλλά μόνο του το Ηνωμένο Βασίλειο ω μεμονωμένη χώρα έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή, δηλαδή είναι σχετικά μικρή έναντι του Ηνωμένου Βασιλείου, ε, έναντι τη Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 ω σύνολο, δηλαδή που έχει πενταπλάσιο ΑΕΠ. Του του το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει χώρα πλούσια με γεωγραφική εγκύτητα βέβαια στην Ευρώπη των 27. Τα μέσα αυτά νούμερα που βλέπετε έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για ορισμένες χώρες και τομείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις οποίες είναι κύριος εταίρος το Ηνωμένο Βασίλειο, περιοχές και τομείς που θα παρουσιάσουν σημαντικά, θα υποστούν σημαντικά πλήγματα από το Brexit. Θα τα δούμε σε λίγο. Ε, συγκεκριμένα οι στατιστικές του εμπορίου τώρα. Μεθοδολογικό, μεθοδολογική επισήμανση. Καταρχάς τα νούμερα που βλέπετε εδώ, που σας παρουσιάζουμε, που έχουμε στην έκθεση, είναι μέσα τιμές της περίοδου 2013-2015. Δηλαδή προσπαθούμε την ανάλυση μας να τη σε, έναν, ε, ε, σε μια εικόνα μέσου όρου ε, κράτους, έτους, συγγνώμη, από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάποιου συγκεκριμένου έτου. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι διμερεί εμπορικέ συναλλαγέ μεταξύ των 27 των κρατών μελών και του Ηνωμένου Βασιλείου είναι γύρω στα 353 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως Μικρό κομμάτι είναι τα γεωργικά, περί το 11% και αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν υπάρξουν συνέπειες στον τομέα της γεωργίας, οι μικροσυνέπειες ε, θα, έχουν περισσότερο, θα εξαρτώνται περισσότερο από αυτά που συμβαίνουν στον παρασκευαστικό τομέα παρά στην παραγωγή. Ε, το εμπορικό συζύγιο βλέπουμε εδώ ότι είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 τόσο στην Παρασκευή όσο και στον ε, γεωργικό τομέα τροφίμων. Έχει σημαντικό ρόλο στις εξαγωγές γεωργικών και τροφίμων του Ηνωμένου Βασιλείου με 9% του συνόλου των εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27 και επίσης εδώ και για λόγους συντομίας θα εστιαστούμε στο χώρο των εξαγωγών, αλλά βέβαια βλέπετε τις λεπτομέρειες στην έκθεσή μας με τα αριθμητικά στοιχεία ε, τα πιο λεπτομερή και μπορούμε να τα συζητήσουμε στη συνέχεια με τις ερωτήσεις. Και το ζήτημα είναι ποιοι είναι οι κύριοι εξαγωγείς, οι κύριοι τομείς που εξάγονται προς το Ηνωμένο Βασίλειο, δηλαδή ποιοι είναι αυτοί οι τομείς και οι εξαγωγές που μπορεί να επηρεαστούν περισσότερο. Βλέπετε εδώ στον πίνακα τους κύριους τομείς εξαγωγών προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εδώ έχουμε για λόγους συνέπειας με το δεύτερο κομμάτι της μελέτης χρησιμοποίηση την ταξινόμηση της βάσης δεδομένων GTAP όπως βλέπετε και έτσι βλέπετε ότι το κύριο εξαγώγημο προϊόν είναι τα τρόφιμα. Υπάρχουν κάποια λυπή τομείς, αλλά κυρίως έχουμε ε, προϊόντα κρέατος, κατεργασμένα προϊόντα όπως μπισκότα κτλ. 17 δισεκατομμύρια συνολικά οι εξαγωγές το χρόνο. Στην πρώτη κατηγορία και έχουμε και το κρέας και λοιπά προϊόντα, γαλακτοκομικά και βόλιο περί τα 11 δις στις εξαγωγές μεγαλύτερες από την, ε, οι εξαγωγές ε, των ποτών και των προϊόντων καπνού που ανέρχονται σε 7 δισεκατομμύρια. Εξαγωγής είναι η Γερμανία, η Γαλλία, 100 χώρες και η Ιρλανδία και στον επόμενο πίνακα και τα επόμενα στοιχεία που επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι ακόμη και αν πάρουμε, αν λάβουμε υπόψη όλους τους τομείς της γεωργίας και των τροφίμων και όλους εξαγωγής, ανάμεικτα πάλι παραμένουν ε, κατά σειρά όγκων ε, ω κύριοι εξαγωγή σε κάτω χώρε η Γαλλία, η Ιρλανδία, η Γερμανία και στην βέβαια ακολουθούν η Ισπανία, η Ιταλία, το Βέλγιο, η Δανία και ούτω καθεξής. Παραμένει δηλαδή αναλογία. Αυτό που βλέπουμε ως σημαντικό με τα κόκκινα είναι το 6% μερίδιο Ιρλανδικών εξαγωγών σε τρόφιμα προς το Ηνωμένο Βασίλειο το τρόφιμα και γεωργικά, πολύ μεγάλο, το πολύ μεγαλύτερο ε, ποσό από ό,τι βλέπουμε για άλλες χώρες που έχουν ποσοστό περί τα 1% πέραν της αξίας. Σημαντικό είναι και το θέμα της προστασίας των ε, ε, εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το Brexit. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει βέβαια τελωνιακό δασμολόγιο για τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά υπάρχουν μη δασμολογικά μέτρα που δεν στοχεύουν ιδιαίτερα το εμπόριο ή τις εξαγωγές, αλλά μπορεί να φέρουν συνέπειες, οι οποίες δεν είναι αμελητές, αντίων και επιπλέον Ίσως χρειαστούν, ε, χρειαστεί προσαρμογή σε κάποιες απαιτήσει σήμανσης, γεωγραφική προέλευση και το καθεξής που μπορεί να επηρεάσουν το εμπόριο, συγκρινόμενο πάντα με τα όσα συμβαίνουν στις εσωτερικές αγορές. Οι μη δασμολογικές λοιπόν, τα μη δασμολογικά μέτρα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι τα κόκκινα με μέσο όρο 18% ισοδύναμο αξία-αξία, ad valorem equivalent, που είναι η αξία δασμού με τις ίδιες συνέπειες με τα μη δασμολογικά μέτρα. Σαν να υπήρχε δηλαδή ο δασμός. Στο γράφημα αυτό βλέπουμε ότι μετά το Brexit και χωρίς συμφωνία εμπορική η προστασία στις εμπορικές συναλλαγές θα παρουσιάσει αύξηση. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στις δύο στήλες σε κάθε κομμάτι του πίνακα. Ε, θα μπουν δασμοί καταρχάς από 0 ε, στην αξία πλέον ευνοωμένου κράτους ε, του ΠΟΕ στο 8% και τα μη δασμολογικά μέτρα επίσης μπορεί να παρουσιάσουν αυξημένη περιοριστικότητα όταν το Ηνωμένο Βασίλειο ή τα 27 κράτη-μέλη αρχίσουν να εισάγουν νέες νομοθεσίες, οι οποίες σιγά σιγά θα αποκλίνουν. Θεωρούμε ότι το 2018 θα έχουμε ένα 20% περισσότερο, μάλλον το 30% πρέπει να είναι η ομιλήτρια, περισσότερο από ότι ε, έχουμε τώρα σε επιβάρυνση με δασμολογική. Οι τομείς που, που θα έχουν τη μεγαλύτερη προστασία είναι οι τομείς με, τη μεγαλύτερη, ε, με τους μεγαλύτερους εμπορικούς όγκους. Γαλακτοκομικά, προϊόντα κρέατος, βόιο, Εκεί θα δούμε τις μεγαλύτερες, ε, το μεγαλύτερο αντίκτυπο. Και ο τελευταίος πίνακας που θα σας αναλύσω είναι αυτός που βλέπετε, όπου αναλύονται οι πληροφορίες αφενός των εμπορικών αξιών, αφετέρου της εμπορικής προστασίας με τους ίδιους τομείς, πάλι με την προηγούμενη διαφάνεια, ταξινομημένου όμως αυτή τη φορά ανάλογα με τον όγκο του εμπορίου, την αξία καλύτερα την εμπορική, πολλαπλασιαζόμενη επί το ποσοστό προστασίας. Και εδώ το κύριο μήνυμα είναι ότι οι τρεις τομείς σε χρώμα πορτοκαλί πλέον παίρνουν ακόμη μεγαλύτερα ποσοστά από ό,τι πριν δηλαδή τα γαλακτοκομικά και τα προϊόντα κρέατος ανεβαίνουν πιο ψηλά από τα αλκοολούχα και τα ε, προϊόντα καπνού. Άρα βλέπουμε μεγαλύτερη διαφορά στους δύο αυτούς τομείς και για τους εξαγωγείς που είναι κυρίως οι κάτω χώρες και η Ιρλανδία. Και θα σας εξηγήσουμε σε λίγο ότι ο απλός δείκτης ε, που έχουμε χρησιμοποιήσει είναι α, αξιόπιστος και δίνει την γενική εικόνα για το ε, εμπόριο, αλλά με την εξήγηση που ο συνάδελφος σε λίγο θα δείτε και την, ε, τη συνέπειες σε μετατόπιση εμπορίου και παραγωγής. Σας ευχαριστώ. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα τα εμπορικά δεδομένα για να εφαρμόσουμε διάφορα μοντέλα μετά το Brexit. Χρησιμοποίησαμε το μοντέλο Mirage, το οποίο αναπτύξαμε. Δεν θα σας απασχολήσω με τις ε, λεπτομέρειες. Βασικά έχουμε ένα σενάριο στο οποίο τα πράγματα θα συνεχίσουν όπως πριν, δηλαδή ε, τι θα γινόταν εάν το Ηνωμένο Βασίλειο παρέμενε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκέρναμε αυτή την κατάσταση με την κατάσταση μετά το Brexit όπου οι δασμοί έχουν αυξηθεί ε, σε ένα καθεστώς ε, ΠΟΕ μάλλον ευνοούμενο κράτους ε, και βεβαίως στην περίπτωση στην οποία έχουν αυξηθεί οι δασμοί όπως ανέφερε ήδη η Σεσίλια. Τα δεδομένα είναι συνεπή και στις δύο περιπτώσεις. Λοιπόν, ε, και έχουμε και το σενάριο Brexit χωρίς εμπορική συμφωνία. Πρώτα απ' όλα λοιπόν έχουμε τα αποτελέσματα στο εμπόριο, αν δούμε το εμπόριο προσπαθούμε εκεί πέρα να κατατάξουμε τους κλάδους και τις χώρες ανάλογα με, τον, με το μέγεθος του αντικτύπου και καταλήξαμε στα ίδια περίπου συμπεράσματα με την Σicilία, δηλαδή βασικά θα είχαμε τεράστια μείωση του εμπορίου, κατά μέσο όρο 62% λιγότερες ε, εξαγωγές από τις 27 προς το Ηνωμένο Βασίλειο και κάποιοι κλάδοι ε, από πλευρά μεγέθου επηρεάζονται περισσότερο από άλλους. Ε, δηλαδή οι λυπή κλάδοι τροφίμων, ζωοτροφές, ε, ζυμαρικά κτλ. Και επίσης ε, τα λευκά κρέατα και τα γαλακτοκομικά. Αλλά αυτό το οποίο είναι πιο ενδιαφέρον είναι ότι για κάποιους συγκεκριμένους κλάδους ε, το εμπόριο σχεδόν καταραίει με πάνω από 90% μείωση. Δηλαδή λευκό κρέας και γαλακτοκομικά αλλά και κόκκινο κρέας και σάκχαρα Εκεί πέρα λοιπόν αυτοί οι τομείς κινδυνεύουν αν υπάρξει Brexit χωρίς εμπορική συμφωνία. Όσον αφορά τις ε, περιφέρειες ε, τώρα, από τις 27 στο, προς το Ηνωμένο Βασίλειο, τις εξαγωγές, έχουμε αυτές τις διαφορές στις χώρες. Οι χώρες οι οποίες επηρεάζονται περισσότερο από πλευράς μεγέθους είναι η μεγαλύτερη εξαγωγή προς το Ηνωμένο Βασίλειο, δηλαδή Ολλανδία, Ιρλανδία και Γαλλία. Αλλά ο σχετικός αντίκτυπος μας λέει πως υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες μπορούν να επηρεαστούν πάρα πολύ όταν μιλάμε για το εμπόριο, ειδικά η Ιρλανδία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μια μείωση ως και 70% των αγροτικών εξαγωγών προς το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και οι υπόλοιποι 27 που δεν αναφέρονται εδώ και η Πολωνία και από την άλλη υπάρχουν κάποιοι κλάδοι, ακόμα και αν είναι μεγάλη εξαγωγή προ το Ηνωμένο Βασίλειο, θα μπορούσαν να ε, είναι σε καλύτερη μοίρα τους άλλους, δηλαδή Γαλλία, Σουηδία και Ισπανία αντιμετωπίζουν μία μείωση 50% και κάτω στο εμπόριο. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες διαφορές. Ο αντίκτυπος λοιπόν στο εμπόριο είναι αυτά τα οποία μας λένε τα δεδομένα. Οι χώρες οι οποίες θα επηρεαστούν από πλευράς όγκου είναι η μεγαλύτερη εξαγωγή, Αλλά αν θέλουμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα υπάρχουν διαφορετικοί παράγοντες που επηρεάζουν. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι εξαγωγές προς το Βασίλειο θα μειωθούν και αυτό βέβαια σημαίνει μείωση της οικονομικής δραστηριότητας ε, στον γεωργικό τομέα. Βλέπουμε εδώ πέρα τις ροζ στήλες ε, που ε, κτίθενται λιγότερο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες και ειδικά το εμπόριο εντός της Ένωσης το οποίο θα αυξηθεί. Γιατί, γιατί η παραγωγή της Ένωσης θα ωφεληθούν από μια νέα προστασία που θα είναι οι δασμοί ε, και μη δασμολογικά μέτρα, άρα θα γίνουν πιο ανταγωνιστικοί από το Ηνωμένο Βασίλειο στην εσωτερική τους αγορά και στην αγορά των άλλων 27. Είναι το μπλε και το μαύρο μέρος της στήλη. Βλέπετε ότι σε κάθε χώρα θα υπάρξει αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας μετά τον Brexit για να εξυπηρεθεί η εσωτερική αγορά και η κοινοτική αγορά, αλλά συνολικά δεν αντισταθμίζει τις απώλειες ε, της αγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου. Αλλά είναι κάπως πιο περίπλοκα τα πράγματα από το να κοιτάμε απλώ το εμπόριο. Και τέλος, είναι οριακό, αλλά θα υπάρξει και κάποια αύξηση της ε, σχετικής ανταγωνιστικότητας ε, στον υπόλοιπο κόσμο για τα γεωργικά προϊόντα της Ένωσης και αυτό γιατί η Βρετανία θα χάσει μέρος της ανταγωνιστικότητάς της γιατί εξαρτάται από την ενδιάμεση κατανάλωση της Ένωσης ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ένα εμπορικό μπλοκ χωρίς δασμούς άρα στην πλευρά των εξαγωγών η σχετική ανταγωνιστικότητα της Ένωσης θα είναι καλύτερη σε σχέση με αυτήν της Βρετανίας. Τέλος, ε, δύο χώρες πραγματικά ξεχωρίζουν εδώ, η Ιρλανδία και η Ολλανδία. Πρώτα γιατί αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη μείωση οικονομική δραστηριότητα ε, και γιατί δεν ωφελούνται από το φαινόμενο αυτό της αύξησης ανταγωνιστικότητας. Και οι χώρες αυτές πραγματικά εξαρτώνται από προϊόντα του Ηνωμένου Βασιλείου, ενδιάμεσα προϊόντα, κατά το οποίο σημαίνει ότι η ανταγωνιστικότητα την οποία θα κέρδιζαν από την προστασία χάνεται γιατί αντιμετωπίζουν υψηλότερο κόστος όταν εισάγουν τα ενδιάμεσα προϊόντα. Οπότε για να πάμε λίγο παραπέρα σε περισσότερες λεπτομέρειες βεβαίως η κατάσταση διαφέρει από τον ένα κλάδο και τη μία χώρα στην άλλη ο χάρτης εδώ σας δείχνει ότι κατά μέσο όρο οι κλάδοι που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι διάφοροι σε κάθε χώρα, π.χ. από γατοτροφές, κιλοτροφές μέχρι κόκκινα κρέατα κτλ. Και κάποιοι κινδυνεύουν ιδιαίτερα, φρούτο-λαχανικά στην Ισπανία ή χοιρινό και πουλερικά στην Ολλανδία. Αυτοί θα επηρεαστούν πάρα πολύ αρνητικά και ενδιαφέρον από την άλλη πλευρά έχουμε κάποιους κλάδους, ε, ελάχιστες σε κάποιες χώρες, που θα ωφεληθούν από το Brexit γιατί τα προϊόντα τους θα υποκαταστήσουν ε, τα βρετανικά προϊόντα στην Ένωση. Π.χ. ο τομέα των βοηδών στην Γαλλία ή το, τα σιτηρά και το στάρι συγκεκριμένα της Ισπανίας. Ε, μιλάμε δηλαδή για υποκατάσταση ε, βρετανικών προϊόντων ή ενδιάμεσα προϊόντα. Για να έχουμε λοιπόν μια γενικότερη άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν δείτε την προστιθέμενη αξία στον τομέα των γεωργικό και των τροφίμων υπάρχουν δύο χώρες, δύο ομάδες χωρών. Η πρώτη ουσιαστικά είναι η Ιρλανδία, η οποία επηρεάζεται περισσότερο από όλους με 16% μείωση στον ε, αγροτοδιατροφικό τομέα. Αυτό τονίζουμε στη μελέτη. Οι άλλες χώρες επηρεάζονται λιγότερο. Το Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία ε, επίσης ε, θα υποφέρουν ε, περισσότερο. Και τέλος, αυτό το οποίο είναι ενδιαφέρον είναι ότι η Βρετανία εδώ εμφανίζεται στο πράσινο, δηλαδή αυτό είναι για να τονίσουμε ότι αν επανέλθουν οι δασμοί, ο Βρετανός παραγωγός επίσης θα έχει μια προστασία στην εσωτερική αγορά, στην εγχώρια του αγορά. Μιλάμε για ένα 2% δεν είναι μεγάλο, αλλά αυτό δείχνουν τα αποτελέσματά μας. Ε, τώρα δεν θα μείνω στα συνολικά αποτελέσματα. Να τονίσω το εξή. Η αύξηση των δασμών σημαίνει αύξηση των τιμών του καταναλωτή οπότε θα εστιάσω μόνο στην αριστερή στήλη. Αυτό το οποίο είναι ενδιαφέρον είναι ότι το αποτέλεσμα αυτό στις τιμές είναι αμεληταίο για όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Δεν επηρεάζεται η τιμή των προϊόντων, σχεδόν κοντά στο μηδέν, αλλά για την Ιρλανδία θα έχει μεγάλο αποτέλεσμα, γιατί η επιβολή δασμών και μη δασμολογικών μέτρων θα μπορούσε να σημάνει 5% συνολική αύξηση στα αγροτοδιατροφικά προϊόντα για τον καταναλωτή. Οπότε, σύντομα τα συμπεράσματα, γιατί απλά επαναλαμβάνω αυτά τα οποία είπα. Βασικό συμπέρασμα είναι ότι ο αντίκτυπος είναι πολύ σημαντικός για την Ιρλανδία και την Ολλανδία και κατά τα λοιπά Υπάρχουν κάποιες προσαρμογές, αλλά το βασικό ζήτημα είναι για αυτές τις δύο χώρες και ειδικότερα την Ιρλανδία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε και περνάμε στις ερωτήσεις. Ο κύριος Άγνιο. Κύριε Άγνιο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, το πιο κρίσιμο τμήμα του Brexit. Οι εμπορικέ σχέσει μετά το Brexit ε, μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα για τα γεωργικά προϊόντα. Και θα είναι χρονοβόρη διαδικασία. Ήδη χάσαμε πολύ χρόνο εξαιτία τη απέτηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση για 100 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν ουρανοκατέβατα εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση ω απέτηση. Και φυσικά δεν μα αρέσει, είναι λογικό νομίζω και όσο ε, συζητούνται αυτά χάνεται πολύτιμος χρόνος και ε, η παραγωγή και η γεωργία από κάποιες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουν σωστές ε, συμφωνίες εμπορικές. Η Γαλλία, η Ιρλανδία, οι κατοχώρες, η Ισπανία θέλουν να επικρατήσει κοινή λογική. Οι γεωργοί τους το απαιτούν για να ομαλοποιηθούν οι μεταγενέστερες εμπορικές σχέσεις με τον Ηνωμένο Βασίλειο. Και δεν φανταζόμουν ε, ότι τόσες πολλές ε, ε, γατό και σκυλοτροφές στέλνονται από τη Γαλλία προς το Ηνωμένο Βασίλειο ή από την Ιρλανδία. Θα ήθελε η παραγωγή να κάνουν να ασκήσουν πιέσεις για διμερείς ίσως συμφωνίες μεταξύ αυτών των χωρών. Αφήστε τι λέει ο Γιούνκερ και ο Μπαρνιέ και η παρελκυστική του τακτική. Εμείς θέλουμε εμπόριο. Επίσης, ε, για την ε, κανονιστική απόκληση, ε, υποτίθεται ότι όταν κάποια προϊόντα εισέρχονται στην αγορά θα πρέπει να πληρούνται οι προδιαγράφεις και κανόνες. Κι όμως από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία οι κτηνοτρόφοι στέλνουν πρόβιο κρέας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να πληρούνται οι ε, διατάξεις για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση των ε, ζώων, ενώ απαιτείται από το Ηνωμένο Βασίλειο να τηρήσει τέτοιου είδους προδιαγραφές και κανόνες. Νομίζω ότι το θέμα του κανονιστικού αποκλεισμού δεν είναι τόσο σοβαρό όσο το παρουσιάζεται. Ευχαριστώ, κύριο Σαντριέ. Σας ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Το κύριο ερωτηματικό, και διορθώστε με κάνω λάθος, είναι ε, ποιες θα είναι οι εμπορικέ συμφωνίε που θα συνάψει το Ηνωμένο Βασίλειο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο είναι τα πιθανά σενάρια. Ή θα παραμείνει στην ισχύουσα Τελωνιακή Ένωση, ένα σενάριο που προδιαγράφεται, το αναφέρατε, ή θα δημιουργήσει ζώνε ελεύθερων συναλλαγών με τι 27 χώρε μέλη. Ανάλογα με το ποιο σενάριο θα επιλέξουμε, οι επιπτώσει είναι πολύ διαφορετικέ. Θα μπορούσατε να μα αναπτύξετε πιο διεξοδικά. Επίση, ποια στοιχεία θα επηρεάσουν τι ήδη Υπάρχουν συμφωνίες. Γιατί το Brexit τέθη αναφιβόλο και πολλές άλλες ισχύουσες ε, συμφωνίες, είτε ελεύθερο εμπορίου, ε, εκεί βέβαια το γεωργικό τμήμα μπορεί να είναι αμεληταίο, αλλά έχουμε και άμεση συνέπειες από τις επιλογές του Ηνωμένου Βασιλείου και το πώς θα επηρεάσουν αυτές οι επιλογές τις ισχύουσες ε, συμφωνίες, εμπορικές συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών. Ευχαριστώ κύριο Ντόρφμαν. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστώ για τη μελέτη. Έχω κανένα δύο ερωτήσεις. Το Ενωμένο Βασίλειο εισάγει αυτά τα προϊόντα, κρέας και τα Έχω κάνει λοιπόν, ε, έχω την εξής ερώτηση. Εάν δεν κάνει τις εισαγωγές, έχετε κάνει μία προσωμείωση σε σχέση με τις ε, εισαγωγέ του Ρωμένου Βασίλου και τι εμπορικέ συναλλαγέ σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο, πώ θα επηρεαστούν οι συναλλαγέ με τον Καναδά, τι Ηνωμένε Πολιτείε ε, τα λοιπά Θα πρέπει να γίνει μια προσαρμογή ασφαλώ στου ε, κανόνε του ΠΟΕ ή συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών για προϊόντα τα οποία τώρα εξάγονται στον υπόλοιπο κόσμο ως προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μετά θα πρέπει να γίνει μια προσαρμογή. Έχετε κάνει αυτή την προσωμείωση και δεύτερον, Έχετε δει μία ανάλυση στους επιμέρους τομείς της, ε, των συνεπειών για προϊόντα που εξάγει το Ηνωμένο Βασίλειο, Φερρυπίν, ε, το ουίσκι που είναι πολύ μεγάλος ε, τομέας. Και βέβαια φαντάζομαι ότι και οι εξαγωγές του προς την Ευρωπαϊκή Ένωση θα δουν ένα δυσμενή αντίκτυπο αλλά και η ανάγκη σε προσαρμογή του κανόνας του ΠΟΕ θα φέρει περισσότερες δυσκολίες. Έχετε, κάνει τους υπολογισμούς. Κύριος Φλάναγκαν, βεβαίως, αν χρειαστεί να επιστρέψουμε στην εισαγωγή κανόνων του ΠΟΕ θα είναι πολύ δυσμενής η συνέπειες για την Ιρλανδία και με ικανοποίηση διαπιστώνω ότι κάποιοι βουλευτές εδώ αναφέρονται στον όρο της αλληλεγγύης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Μπαρνιέ θα έπρεπε λοιπόν, αν είναι έτσι τα πράγματα, να λάβει υπόψη ότι η Ιρλανδία είναι αυτή η οποία θα υποφέρει περισσότερο. Άκουσα από το Προεδρείο να λέγεται πως ε, η Βρετανία δεν θα πρέπει να επιλέξει μια κατάσταση η οποία θα οδηγήσει σε επιδείνωση των συνθήκων. Βεβαίως και μπράβο σας, αλλά Ταυτόχρονα ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενοχλημένη με τον Ενωμένο Βασίλειο και το Ενωμένο Βασίλειο ενοχλημένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σαν να τσακώνεται ένα ζευγάρι για το ποιο θα πάρει την επιμέλεια των παιδιών ύστερα από ένα διαζύγιο. Εμεί όμω είμαστε αυτοί που θα υποφέρουμε περισσότερο. Αν λοιπόν υπάρχει αλληλεγγύη, αν και δεν το είδα αυτό, ούτε ω προ τα χρέη στις τράπεζ, των τραπεζών, ούτε όταν ε, κλήθησαν οι Έλληνε να πληρώσουν, ο ελληνικός λαός να πληρώσει λογαριασμό αυτών που τους έχουν καταστρέψει. Ε, ωστόσο, εάν υπήρχε αυτή η ελεγγύη, επανέρχομαι, θα έπρεπε με τον, για το Ηνωμένο Βασίλειο να παραμείνει κάποια μορφή τελωνιακής ένωσης, εάν παρέμεναν και οι δύο πλευρέ αρκετά λογικέ, αν και δεν βλέπω αυτό να συμβαίνει. Βλέπω καθένα να προσπαθεί να κερδίσει από ένα πόντο ε, κάθε φορά για να δείξει ότι την έφερε στον άλλον. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε κάποιες διαφορετικέ εξελίξει. Ευχαριστώ πολύ, Κάρτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε και θα συνεχίσω στα όσα επεσήμανα νωρίτερα. Ευπρόσδεκτη και αυτή η έκθεση δίνει πολύ ξεκάθαρα την εικόνα και αναφέρεται, όπως είπα και εγώ νωρίτερα, στις συνέπειες για τους Ιρλανδούς γεωργούς από το Brexit και νομίζω μπορεί να αποτελέσει ε, και αφύπνιση για κάποιους που θεωρούν ότι θα τους συνέφερε, κάποιους γεωργούς που θεωρούν ότι θα του συνέφερε το Brexit. Βεβαίως η Βόρεια Ιρλανδία δεν έχει συγκεκριμένα στοιχεία, δεν αναφέρονται συγκεκριμένα στοιχεία για, την Ιρλανδία, για τη Βόρεια Ιρλανδία στι μελέτες σας και νομίζω ότι θα είναι πολύ πιο σοβαρές οι συνέπειες ε, ε, για τους γεωργούς της βόρεια Ιρλανδίας από ό,τι για τους υπόλοιπους. Υπάρχει λύση όμως, υπάρχει λύση και η λύση θα έπρεπε να είναι να παραμείνει στην Τελωνιακή Ένωση ολόκληρη η Ιρλανδία το βόρειο και το νότιο τμήμα ε, στην ενιαία αγορά, γιατί κάθε άλλη λύση θα ήταν καταστροφική. Είτε πρόκειται για την ασφάλεια των τροφίμων και τη σχετική νομοθεσία, είτε για την ε, είτε για άλλους όρους συνοχής ε, θα ήταν καταστροφικές οι συνέπειες αν παρέμενε στο, στο Ηνωμένο Βασίλειο ως αγορά η Βόρεια Ιρλανδία. Εάν λοιπόν θέλουν οι Βρετανοί πραγματικά να προχωρήσουν σε μια απρόσκοπτη και ομαλή έξοδο χωρίς να παραβλαφθεί και το σύστημα των ανοιχτών σύνορων μεταξύ Δημοκρατίας Ιρλανδίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουν και νομίζω ότι έτσι μπορούν να λυθούν όλα τα προβλήματα με μία και μόνη απόφαση. Εάν δεν το πράξουν όμως αυτό και αν αποφασίσουν ότι αποχωρούν και αρχίζουν να κοπηλατούν μόνοι τους, τότε θα πρέπει να, κάνουμε, να βρούμε λύσεις διμερώς. Και όταν, αρχίσουν, ε, όταν πλέον έχουν ολοκληρωθεί οι ε, διαδικασίες αναγνώρισης διμερώς των προϊόντων μεταξύ Βόρειας Ιρλανδίας και ε, Δημοκρατίας Ιρλανδίας, τότε θα έχει έρθει η ώρα για την ε, επαλήθευση της πραγματικής αλληλεγγύης από πλευράς της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, δηλαδή αν θέλει πράγματι το σεβασμό της Συμφωνίας Μεγάλης Παρασκευής και όλης αυτής της πορείας για την ειρήνευση στην ίνεση της Ιρλανδίας των τελευταίων 20 ετών, της προστασίας της ε, οικονομίας του γεωργικού τομέα σε ολόκληρη την ίσο της Ιρλανδίας, συμπεριλαμβανομένου και του βόρειου τμήματος. Εκεί θα γίνει η δοκιμασία. Ευχαριστώ κύριε Μαγκίνες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω λίγες ερωτήσεις σε σχέση με τα βασικά σας πορίσματα. Είπατε ότι μερικές εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταρρεύσουν πλήρως και μας τις απαριθμίσατε. Σήμερα, όσο εμείς συζητούμε, γίνονται κάποιες διαπραγματεύσεις, αλλά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε, αν ε, καταλήξουμε σε μη, συμφωνία, πώς θα ε, καλύψει το κενό ή πώς θα γεμίσει τα ράφια του σούπερ μάρκετ το Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί μέχρι στιγμής ε, τα τρόφιμα παραδίδονται εγκαίρως, δεν υπάρχουν ελλείψεις ε, και πληρούνται οι κανόνες και οι προδιαγραφές και για τους καταναλωτές και για τους λιανεμπόρους. Ε, μιλήσατε όμως για ένα σενάριο πλήρους κατάρρευσης κάποιων εξαγωγών ορισμένων προϊόντων. Δεν μπορώ καν να το διανοηθώ. Ε, κάποιες χώρες όπως και η πατρίδα μου η Ιρλανδία θα επηρεαστούν πολύ πιο σοβαρά από ένα τέτοιο σενάριο και ε, ουσιαστικά επιβεβαιώσετε αυτά που ήδη γνωρίζουμε. Αν όμως είχαμε μια μετατόπιση ε, του βοήου κρέατος και του τυριού τσένταρ, κυρίως εκτός της αγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου, λόγω σκληρού Brexit, αυτό δεν είναι πρόβλημα μόνο για την Ιρλανδία, γιατί τα προϊόντα αυτά πρέπει κάπου να αναζητήσουν αγορές και θα τις βρουν είτε στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση και ίσως και με χαμηλότερες τιμές ή σε αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να μας αναπτύξετε κάπως πιο δελεχώς αυτό το σημείο. Γιατί σίγουρα είμαστε κόκκινοι στο χάρτη και ξέρουμε ότι είμαστε στη ζώνη κινδύνου. Αλλά αυτό ο κίνδυνο δεν θα παραμείνει εντό τη Ιρλανδική επικράτεια. Επίση, έχουμε το επιπρόσθετο πρόβλημα. Πολλέ πρώτε ύλε στην ίσο τη Ιρλανδία είναι ευρωπαϊκές. Οπότε δεν κάνουμε διάκριση ε, πώς παράγεται ε, το γάλα, αν είναι βόρειο των σύνορων ή αλλού. Ή όπως ε, θα διαπιστώσει και ο κύριος Νίκολσον, κάποιες αγελάδες μπορεί να βοσκούν στην μια πλευρά των σύνορων, αλλά να τις αρμέγουν στην άλλη πλευρά των σύνορων. Οπότε όλα αυτά θα επηρεαστούν ανάλογα με το σενάριο που θα επιλέξουμε. Και η ιδέα του να μην υπάρχει σύνορο, γιατί αυτό σίγουρα είναι ο στόχο, μη τι άλλο, τη Ιρλανδία. Και το, το συμπέρασμα είναι, όπω σα επαναλαμβάνω συχνά, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να παραμείνει στην Τελωνιακή Ένωση. Ευχαριστώ, κύριο Νίκολσον. Ευχαριστώ. Οποιοδήποτε γνωρίζει κάτι για το θέμα αυτό ε, καταλαβαίνει ότι αν ε, πάνε τα πράγματα στραβά θα γυρίσουμε ε, στους καρόνες του ΠΟΕ και αυτό θα είναι φιάλτης για όλους. Όλοι θα βρεθούμε χαμένοι. Δεν θα υπάρξει κανένας κερδισμένος από μια τέτοια λύση. Ε, κύριε Μακάρθη, ε, έχετε κάνει πολλά ανακοινωθέντα τύπου, αλλά εκεί περιορίζεται και δεν κάνετε προτάσεις για να επιληθούν τα προβλήματα. Η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι το εμπόριο βρίσκεται στο κέντρο της λύσης και δεν μπορούμε να λύσουμε ένα πρόβλημα που καλούμαστε να επιλύσουμε αν δεν ασχοληθούμε και με την εμπορική πτυχή που βρίσκεται στο επίκεντρο. Κύριε Κάρθη, από ό,τι κατάλαβα, το 80% των αγροδιατροφικών της ε, Ιρλανδίας διοχετεύονται απευθεία στη Βρετανική αγορά. Και αυτό δεν ε, υπάρχει πλέον, δεν υπάγεται στο, στον ΠΟΕ. Τώρα θα δημιουργηθεί πρόβλημα στη δημοκρατία της Ελλαδίας που θα εμπίπτουν αμέσω ε, στις κανόνες του ΠΟΕ αν δεν υλοποιηθεί η συμφωνία. Και όλοι μας λένε ότι θα πρέπει να σκεφτόμαστε διορατικά και πρωτότυπα και Μιλούμε για την Τελωνιακή Ένωση και την εσωτερική αγορά. Η Τελωνιακή Ένωση όμως και η εσωτερική αγορά δεν, ήταν, δεν υπήρχαν από την αρχή. Δημιουργήθηκαν, η Τελωνική Ένωση δημιουργήθηκε λόγω της εσωτερικής αγοράς. Δεν είναι λοιπόν λογικό και εφικτό αν φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο να έχουμε μια νέα Τελωνιακή Ένωση και νέα συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου. Κάτι τέτοιο θα επίλυε πολλά προβλήματα. Και μη λέτε ότι η Τελωνιακή Ένωση δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτό το αμφισβητώ θα πρέπει να είμαστε πιο διορατικοί και αν θέλουμε να είμαστε ευρηματικοί και δημιουργικοί και πραγματικά να βρούμε λύση για να λύσουμε τα προβλήματα, θα πρέπει να ανοίξουμε τους ορίζοντάς μας και να σκεφτούμε και τέτοιες λύσεις. Ο κύριος Μπάνων. Ναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρά το ότι ψήφισα να παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο, θεωρώ ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε την θετική πτυχή σε όλα αυτά. Βεβαίω, ε, μάθαμε σήμερα πώς δουλεύει το εμπόριο εντός της Ένωσης και πόσο ταξιδεύουν τα τρόφιμα. Ε, το γράφημα σελίδα 35 είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί η Ολλανδία και η Ιρλανδία ε, έχουν και θέμα βεβαίως γεωγραφικής εγκύτητας με το Ηνωμένο Βασίλειο, γι' αυτό πλήττονται περισσότερο. Δεν προξενεί εκπλήξη ότι οι πιο κοντινέ χώρε εμπορεύονται περισσότερο με το Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με τι πιο μακρινέ. Και από τη σκοπιά του Ηνωμένου Βασιλείου, αν εμπορευτούμε λιγότερο με την Ευρωπαϊκή Ένωση και περισσότερο με τον υπόλοιπο κόσμο, θεωρητικά ίσω έχουμε φθηνότερα τρόφιμα, αλλά θα αυξηθούν περισσότερο τα μίλια που διανύουν τα τρόφιμα και ο αντίκτυπο στο περιβάλλον και το κλίμα θα είναι μεγάλο. Και αν ψάχνουμε λοιπόν κάποια θετική πτυχή μήπως ε, θα πρέπει να σκεφτούμε και εμείς το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή το θέμα του πόσο μακριά ταξιδεύουν τα τρόφιμα και μήπως να τρώμε και ε, φρουτολαχανικά εποχής όχι όλο το χρόνο και να δούμε διαφορετικά το θέμα των τροφίμων ίσως αυτό να είναι ένα από τα θετικά που θα προκύψουν παρά το ότι βεβαίως η γενικότερη κατάσταση θα είναι άσχημη. Σας ευχαριστώ. Δεν έχουμε άλλους ε, ε, ομιλητές στο κατάλογο, οπότε ένα δεκάλεπτο έχουν ακόμη οι εμπειρογνώμονές μας για να απαντήσουν στις ερωτήσεις, αλλά ούτε λεπτό παραπάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις σας. Να απαντήσω πρώτα για το θέμα της Βόρειας Ελλανδίας. Βεβαίως θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε ακριβώ τις λεπτομέρειες αυτής της ε, περιφέρειας του Ηνωμένου Βασιλείου. Το πρόβλημα είναι ότι αφενός τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιούμε δεν είναι τόσο ακριβή και από την άλλη θέλαμε να εστιάσουμε κυρίως ε, στα υπόλοιπα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί ήδη έχουν υπάρξει αρκετές μελέτες. Μπορείτε να δείτε τη βιβλιογραφία στην μελέτη μας για το τι θα συμβεί στην Βρετανία και τους Βρετανούς ε, αγρότες και ειδικά αυτούς της ε, Βορείου Ιρλανδίας. Οπότε δυστυχώς δεν υπάρχουν κάποια στοιχεία για αυτό το θέμα. Το δεύτερο θέμα το οποίο προέκυψε πολλές φορές είναι το τι μπορούν να κάνουν τα κράτη-μέλη και το Ηνωμένο Βασίλειο για να αποφύγουν αυτήν την κατάσταση. Αυτό το οποίο είδαμε, αλλά δεν ήταν στην μελέτη γιατί δεν μας ζητήθηκε από το Κοινοβούλιο, το οποίο επέμενε για το σενάριο του ΠΟΕ και ήθελε τα αποτελέσματα, τα νούμερα. Προσπαθήσαμε να δούμε το ποια θα ήταν η κατάσταση με μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ένωσης ε, και βεβαίως ε, κομμάτι του αντίκτυπου που ανέφερα ε, εξαφανίζεται, αλλά όχι όλες οι επιπτώσεις γιατί πολλά ζητήματα ε, υπάρχουν και το βασικό θέμα είναι η ρυθμιστική απόκληση και ειδικά τα μεγαλύτερα ε, θέματα και κλάδη. Να αναφέρω ένα πράγμα. Η σύγκριση μεταξύ του των μπλε και των μαύρων στυλών ε, οι στήλε είναι τα διάφορα σενάρια με τις μπλε στήλες δεν υπάρχει ρυθμιστική απόκληση και το Ηνωμένο Βασίλειο τηρεί τους ίδιους κανόνες με την Ένωση και για πολλούς κλάδους έχουμε τον μισό αντίκτυπο στο εμπόριο αλλά για ε, τους κλάδους που επηρεάζονται περισσότερο, λευκά κρέατα, γαλακτοκομικά και κόκκινα κρέατα, βλέπουμε πάλι πλήρη εξαφάνιση του εμπορίου. Γιατί είναι πολύ σημαντική η δασμή, αλλά για άλλους κλάδους ε, το θέμα αυτό της ρυθμιστικής απόκλησης είναι το σημαντικότερο. Αλλά όχι για αυτό το θέμα ίσως. Ναι. Για τον κλιματικό αντίκτυπο και τα μίλια που διασχίζουν τα τρόφιμα υπάρχουν καλά και κακά νέα με αυτές τις ε, περιπτώσεις το καλό είναι ότι λιγότερα αγαθά θα διασχίζουν τη μάχη ε, και για το Ηνωμένο Βασίλειο ίσως ε, ο παγκόσμιος αντίκτυπος, ε, ο συνολικός με συγχωρείτε αντίκτυπος να είναι καλός. Δεν έχω δει τα νούμερα. Θα πρέπει να τα δούμε προσεκτικά πριν βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα. Αλλά δεν είναι σαφές ότι θα είναι κακό για το περιβάλλον και για να έρθω στο θέμα του που πηγαίνουν ε, τα προϊόντα αν δεν θα πηγαίνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχετε δίκιο κυρία Μαγκίνες όταν λέτε ότι πηγαίνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη σε φτηνότερες τιμές. Γι' αυτό έχουμε αυτόν τον αντίκτυπο για τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Εάν, καταναλωτές. δείτε στην τελευταία διαφάνεια στην αριστερή στήλη κάποιοι κλάδοι ευνοούνται, αλλά συνολικά, στο σύνολο όλα τα προϊόντα, όχι μόνο τα κρέατα, για Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία, βλέπετε ότι οι καταναλωτές τους ε, ωφελούνται από τις χαμηλότερες τιμές ε, λόγω του ότι πλεονάζει η παραγωγή κρέατος και λοιπόν προϊόντων. Αλλά ε, δεν είναι ουσιαστικό σε σχέση με τον αρνητικό αντίκτυπο για τους καταναλωτές λόγω των δασμών. Και ε, ξανά και εδώ είναι τελείως διαφορετική η κατάσταση για την Ιρλανδία. Έχετε κάτι να προσθέσετε. Στο θέμα των ε, εμπορικών συμφωνιών με τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι πολύ περίπλοκο. Και θα έλεγα ότι έχει και νομικά περισσότερο χαρακτηριστικά παρά οικονομικά. Κύρια απάντηση που μπορώ να σας δώσω είναι ότι παραμένει τεράστια βεβαιότητα και δεν ξέρουμε τεχνικά τι λύσεις θα βρεθούν. Τι θα συμβεί. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι την κατάσταση πάντως, οι εμπορικές συμφωνίες που αφορούν μόνο αγαθά, αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ω εκ τούτου θα πρέπει να ξεκινήσει εκ νέου η διαπραγμάτευση από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ιδάλω, απλώ ε, εκπνέουν, εξαφανίζονται όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι το μόνο που φαίνεται βέβαιον. Για όλα τα άλλα παραμένει η αβεβαιότητα. Για την ε, προσωμείωση τώρα και την έκθεσή μα. δεν αλλάξαμε τίποτα και άρα το Ηνωμένο Βασίλειο διατηρεί τους ίδιους δασμούς και την προστασία στο, εμπορικό, στο εμποριό του προς όλες τις χώρες, είτε εισάγει είτε εξάγει. Το, μόνο, το ίδιο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο αλλάζουν οι δασμοί και η εμπορική προστασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου. Άρα απομονώνουμε τις συνέπειες της και σχέση, αλλά πολλά άλλα μπορούν να συμβούν. Ε, ένα ολόκληρο πλέγμα δηλαδή σχέσεων μπορεί να εξαρτούνται από αυτό, αλλά είναι βέβαιο. Όπως είπε και ο συνάδελφος. Έχουμε κάνει κάποιες προσωμιώσεις και με διαφορετικά σενάρια. Ίσως θα μπορούσαμε να σας δώσουμε έναν-δύο πίνακες ακόμη γραφήματα. Ποσοστώσεις επίσης στις εμπορικές συναλλαγές. Άλλο ένα τεράστιο και πολύ πολύ αβέβαιο θέμα, όπου πάλι δεν έχουμε συγκεκριμένες υποθέσεις κάνει, για αλλαγές δηλαδή σε δασμολογικά συντελεστές, ε, αλλά είναι πιθανόν ότι θα συμβούν. τα αγαθά που δεν, εξάγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, που δεν θα εξάγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο θα βρούνε κάπου αλλού εναλλακτικέ ε, ε, και σχετικά ερωτήματα. Κάποιες υποθέσεις ή γενικές ιδέες που μπορώ να σας προσφέρω είναι ότι η βαρύτητα έχει πολύ μεγάλη σημασία και στο εμπόριο. Οι εξαγωγές σας λοιπόν θα τίνουν να πάνε, προ... οι εξαγωγές δηλαδή τίνουν να πηγαίνουν στον εγκύτερο και το μεγαλύτερο εταίρο. Και μετά υπάρχουν και υπάρχει και η έννοια της τριβής στο εμπόριο. Δηλαδή αν είσαι κοντά μου θα εξάγω σε σένα μεν, αλλά αν υπάρχει άλλος εταίρος μεγαλύτερος, έστω και πιο μακριά, θα εξάγω προς αυτόν. Αυτή είναι μια κάποια ιδέα που μπορώ να σας δώσω και Επίσης υπάρχουν οι τάσεις, τα προϊόντα που παραδοσιακά εξάγονταν στο Ηνωμένο Βασίλειο να μένουν σε ένα βαθμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα μέρος τους μόνο να βγαίνει εκτός. Αλλά όπως είπα θα μπορούσαμε να είχαμε περιλάβει και άλλα στοιχεία στην έκθεση και άλλες αναλύσεις. Η κυρία Μαγκίνη ζήτησε μισό λεπτό ακόμη μπορείτε να μας απαντήσετε τι θα γίνει με τη διαταραχή στην ε, αλυσίδα προσφοράς, προμήθειας. Ε, μπορεί να μην υπήρχε στη μελέτη, αλλά θα μπορούσατε να το σχολιάσετε. Το θέμα της αλυσίδας ε, νεφοδιασμού καλύπτονται, καλύπτονται στη μελέτη, αλλά όχι αμέσως, εμέσως. Και μάλιστα έχουμε ένα τμήμα που αφορά τις εναλλαγές ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου και τη διασύνδεση των αλυσίδων ε, ανεφοδιασμού. Πάντως την προσωμείωση με το εμπορικό σενάριο, με την επαναφορά των κανόνων του ΠΟΕ, ε, έχουμε και το στοιχείο των αλυσίδων ανεφοδιασμού, αλλά δεν αναφέρονται ρητά σε τέτοιου μοντέλα. Ε, υπάρχουν άλλες μελέτες που δίνουν λεπτομέρειες. Στη δική μας μελέτη είχαμε απλώς τις ε, έμεσες ε, εισρωές, την κατανάλωση των επιχειρήσεων και κατά μέσο όρο την προέλευση. Οπότε πώς οργανώνονται κατά μέσο όρο αυτές οι αλυσίδες ανεφοδιασμού αναχώρα, αλλά όχι ανατομέα. Οπότε τα πιο πρόσφατα μοντέλα αρχίζουν να λαμβάνουν υπόψη και αυτό το στοιχείο των επιμέρους τομέων. Με τέτοιου είδου μοντέλα που είχαμε μέχρι στιγμής δεν ήταν δυνατόν να συμπεριλάβουμε και τέτοια στοιχεία στη μελέτη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θερμά τους εμπειρογνώμονές μας. Αλλαγή τώρα φρουρά. Περνάμε στο, στην επόμενη ομιλία με θέμα τις πιθανές μεταβατικές συμφωνίες για τη Γεωργία υπό το φως των μελλοντικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε το γνωστό γνώριμο στην Επιτροπή μας καθηγητή από το Trinity College του Δουβλίνου, τον κύριο Άλα Μάθιους. Είχαμε τη χαρά να τον φιλοξενήσουμε επανειλημμένο στην Επιτροπή μας. Παρακαλώ κύριε Μάθιους, λάβετε θέση. Έχετε και εσείς 20 λεπτά, ίσως δεν χρειαστείτε βέβαια να τα εξαντλήσετε. Ευχαριστώ, καλημέρα σας. Είχα τη χαρά να σας παρουσιάσω εδώ το τρίτο τμήμα. Η μελέτη μου ήταν αρκετά μακροσκελής και διεξοδική, αλλά νομίζω ότι σε αυτή τη φάση της διαδικασίας ε, οι λεπτομέρειες είναι σημαντικές. Θα σας παρουσιάσω τις αδρές γραμμές της μελέτης και τα βασικά μηνύματα του εγγράφου παρακάπτοντας ε, πολλές λεπτομέρειες και αφήνοντας χρόνο και για τις ερωτήσεις. Σημείο φετηρίας φυσικά είναι γνωστό σε όλους. Η Βρετανίδα Πρωθυπουργό στην ε, ομιλία της ε, στο Λάνκαστερ και στις δηλώσεις που έκανε στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στην ομιλία της στη Φλωρεντία είπε φυσικά ότι το Ηνωμένο Βασίλειο σκοπεύει να αφήσει και την Τελωνιακή Ένωση, να καταλήψει και την εσωτερική, την ενιαία αγορά και ζητά μια φιλόδοξη και τολμηρή συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επισήμανε κάποιε όμω κόκκινε γραμμέ ε, για το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Από πλευρά ε, Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε τι κατευθυντήριε γραμμέ που συμφωνήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Έχουμε μέχρι στιγμής και τα δύο ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τις δικές του κατευθυντήριες γραμμές και το βασικό μήνυμα εκεί είναι ε, μια χώρα που δεν θα είναι μέλος και ε, δεν μπορεί να έχει τις ίδιες υποχρεώσεις ε, με τις ε, υπόλοιπες χώρες μέλη και άρα δεν μπορεί να διεκδικεί και τα ίδια δικαιώματα. Επίσης αναφέρθηκε μια ε, ένα χρονοδιάγραμμα για τις διαπραγματεύσεις ε, και είχαμε και το θερινό ε, συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του περασμένου μήνα που διαπίστωσε την έλλειψη πρόοδου ή την ανεπαρκή πρόοδο στην πρώτη φάση των διαπραγματεύσεων για τα τρία βασικά στοιχεία, την ηθαγένεια, τα δικαιώματα των πολιτών, τις οικονομικές διευθετήσεις και το ζήτημα των Ιρλανδικών σύνορων, του Ιρλανδικού σύνορου. Πάντως δόθηκε το μήνυμα ότι το Συμβούλιο και ο διαπραγματευτής εκ μέρους Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ξεκινήσουν τις ε, εσωτερικές ε, προετοιμασίες για να διαμορφώσουν τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τις μελλοντικές εμπορικές ε, σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και τις μεταβατικές συμφωνίες. Με βάση αυτό λοιπόν το υπόβαθρο ε, αυτό που επιχείρησα στη μελέτη αυτή είναι να εξετάσω τρία πρωταρχικά ζητήματα. Καταρχήν, να εντοπίσω με όλες τις δυνατές λεπτομέρειες ποιες είναι οι εμπορικές συνέπειες της ε, θέσης του Ηνωμένου Βασιλείου και πώς οι μελλοντικές εμπορικές σχέσεις μπορεί να μετριάσουν, και το τονίζω αυτό, να μετριάσουν, γιατί θα πρέπει να ε, αναγνωρίσουμε ότι από τη στιγμή που το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταλήψει την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούμε να έχουμε τις ίδιες ε, οι απρόσκοπτες εμπορικές σχέσεις που έχουμε μέχρι στιγμής. Είναι αδύνατο και αυτό θα πρέπει να το ε, λάβουμε υπόψη. Αλλά μπορούμε να μετριάσουμε μερικές από τις συνέπειες και εξετάζω ε, πιθανότητες για να το κάνουμε. Δεύτερον, ακόμη και αν καταλήξουμε σε συμφωνία στις ε, διαπραγματεύσεις του άρθρου 50 για τους όρους της αποχώρησης και έχουμε μια έφτακτη αποχώρηση, ε, υπάρχει το, η εύλογη ανησυχία να μην προλάβουμε μέχρι το Μάρτιο του 2019 να, να είμαστε έτοιμοι για να εφαρμόσουμε αυτή τη συμφωνία. Οπότε νομίζω ότι και οι δύο πλευρές έχουν ε, αποδεχθεί την ανάγκη κάποιων μεταβατικών ρυθμίσεων. Οι Βρετανοί το λένε περίοδο εφαρμογής, για να αποφύγουμε αυτό το χείλο του κρεμού και θα σας αναλύσω πώς μπορούμε να το αποτρέψουμε αυτό στην πράξη. Και το τρίτο τμήμα της μελέτης αναγνωρίζει ότι είτε θα έχουμε μια κατάσταση έφτακτης αποχώρησης, αλλά τι θα γίνει σε περίπτωση που έχουμε μια άτακτη αποχώρηση, αν να βαγίσουν δηλαδή οι διαπραγματεύσεις, κάτι που είναι και αυτό μια πιθανότητα. Και όπως ανέφεραν και δύο προηγούμενες μελέτες, ε, οι συνέπειες μη συμφωνίας θα είναι αρνητικές για, γενικώς για τους γεωργούς, συγκεκριμένα για τους γεωργούς ε, κάποιων χωρών. Και εγώ αναλύω και τις πιθανότητες που, και δυνατότητες μάλλον που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και επιλογές για να προσπαθήσει να αντισταθμίσει μερικές από αυτές τις ζημίες. Αυτά τα τρία θέματα λοιπόν θα συζητήσουμε. περνάμε στις εμπορικές επιπτώσεις. Ε, σε περίπτωση που έχουμε σκληρό Brexit, που ανέλησαν και οι προηγούμενες μελέτες. Η πρώτη και πιο σημαντική συνέπεια θα είναι η επαναφορά των δασμών στο εμπόριο μεταξύ των 27 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές από το Ηνωμένο Βασίλειο, γνωρίζουμε ότι οι δασμοί που θα επιβληθούν στις ε, βρετανικές εξαγωγές, γιατί ε, μπορείτε να δείτε στο ΤΑΡΙΚ, ε, στον κοινό εξωτερικό δασμό, για μερικά προϊόντα οι δασμοί αυτοί μπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλοί. Τώρα για τους Ευρωπαίους εξαγούς προς το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι ακόμη σαφέ τι επίπεδο δασμών μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο, όταν το Ηνωμένο Βασίλειο γίνει τρίτη χώρα. Το Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε ότι θα επαναφέρει τους δασμούς του ΠΟΕ, δηλαδή τους ανώτατους δασμούς. Δεν θα ξεπεράσει όμως αυτό το ανώτατο όριο που ισχύει. Από τη στιγμή όμως που θα έχει την αυτονομία ε, της εμπορικής του πολιτικής μπορεί να μειώσει αυτούς τους δασμούς. Κάποιες φωνές, όχι στην κυβέρνηση, αλλά ακούγονται κάποιες τομέ εκτός κυβέρνησης του ΕΒ που επιχειρηματολογούν σε περίπτωση που θέλουν να γίνει παγκόσμιο εταίρο του ΕΒ Βασίλειο, να χρειαστεί μονομερό να μειώσει του δασμού των προϊόντων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρουμε λοιπόν γιατί επίπεδο δασμών μιλάμε. Πάντω είναι λογικό να εικάζουμε, όπως είπε και προηγούμενη μελέτη, ότι αρχικά οι δασμοί που θα εφαρμοστούν θα είναι αρχικά τουλάχιστον στο επίπεδο αυτό που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε τρίτες χώρες, δηλαδή υψηλή δασμή στο εμπόριο. Δεύτερο στοιχείο που δεν αφορά μια εμπορική, εμπορικό κόστος, αλλά ε, την απώλεια των ε, προνομιακών, των προτιμησιακών ε, εμπορικών ε, μεταφορών. Και σε... οι τιμές των τροφίμων επηρεάζονται γιατί εφαρμόζονται οι ίδιες ταρίφ, οι ίδιοι δασμοί στις εισαγωγές τρίτων, προϊόντων τρίτων χωρών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όταν οι εξαγωγοί πουλούν στην Ευρωπαϊκή ευρωπαϊκή αγορά έχουν το πλεονέκτημα μιας προτιμησιακής τιμής που είναι υψηλότερη από την παγκόσμια τιμή αγοράς. Και αν διαθέταμε τα προϊόντα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα είχαμε αυτή την προτιμησιακή τιμή την οποία απολαμβάνουμε στην ενωσιακή αγορά. Οπότε θα χάσουμε αυτές τις προτιμησιακές τιμές σε περίπτωση σκληρού exit. Τώρα, αν το Ηνωμένο Βασίλειο ε, μειώσει τους δασμούς ή τους εκμηδενήσει, ε, και στις συμφωνίες αυτές ε, αποφύγουμε τους, ε, δασμολογικού τους δασμολογικούς φραγμούς και πάλι το Ηνωμένο Βασίλειο θα ήταν λιγότερο ελκυστική αγορά αν μείωνε μόνο μονομερός τους δασμούς κάτω από το ισχύον σήμερα επίπεδο. Αυτός είναι ένας τρόπος που η ελκυστικότητα της Βρετανικής αγοράς θα μπορούσε να μειωθεί. Ε, ένα άλλο στοιχείο θα ήταν να έχουμε και δασμούς ε, εξαγωγών προς το Ηνωμένο Βασίλειο στο σενάριο του σκληρού Brexit και εκεί το Ηνωμένο Βασίλειο να διατηρήσει σχετικά υψηλούς ε, δασμούς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά να υπογράψει συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου με ανταγωνιστικούς εξαγωγείς Αυστραλία, Καναδά, χώρες του Μερκοσούρ και ούτω καθεξής ώστε τα επίπεδα τιμών στην Βρετανική αγορά να πέσουν. Σε τέτοια περίπτωση θα έχουμε και υψηλότερου δασμούς για τις εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο και θα είναι και ελκυστικό ε, το Ηνωμένο Βασίλειο η τιμή δηλαδή που ο εξαγωγός ε, θα λάμβανε ακόμη και ξεπεράσει το τείχος θα ήταν χαμηλότερη. Βέβαια είναι λιγότερε αυτέ οι απώλειε από ό,τι πήρε από μία δεκαετία εξαιτία ε, των σταδιακών μεταρρυθμίσεων τη κοινή γεωρική πολιτική και το γεγονό ότι έχουν αυξηθεί οι παγκόσμιε τιμέ τα τελευταία χρόνια. Αλλά για κάποια αγαθά, για κάποια προϊόντα, για βόλιο και κρέα πουλερικών, θα είχαμε σημαντική απώλεια προτιμησιακών τιμών για τον Βρετανό καταναλωτή. Τρίτον, το κόστο του εκτελονισμού Φυσικά το κόστος αυτό μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με κάποιες τελωνιακές συμφωνίες κάθε τύπου, αλλά ακόμη και αν έχουμε ελεύθερα σύνορα, Νορβηγία, Σουηδία, όπως ε, τέτοιο παράδειγμα, ή Γαλλία, Γερμανία απέναντι στην Ελβετία, ακόμη και αν έχουμε τέτοιου είδους σύνορων και πάλι θα υπάρχει έλεγχος τελωνιακός, είτε για λόγους υγειονομικούς, είτε κάποιοι έλεγχοι ταυτότητας Και φυσικά για τα αγροδιατροφικά προϊόντα που φτάνουμε στο, στην τέταρτη συνέπεια θα έχουμε επιπλέον και κόστος ε, κανονιστικής συμμόρφωσης. Γενικώ για τα τρόφιμα ε, μη ζωικής προέλευσης δεν υπάρχει απέτηση ε, για προέγκριση, προπιστοποίηση προκειμένου να γίνουν εισαγωγέ από συγκεκριμένα, να περάσουν από συγκεκριμένα σημεία. Αλλά για τα προϊόντα ζωική προέλευση η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ αυστηρού κανόνε και εκεί μπορεί κανείς να εισάγει τα προϊόντα του ε, σε σημαντικούς πόλους ε, επιθεωρήσω στα σύνορα. Εκεί έχουμε και εργαστήρια και χώρους αποθήκευσης, ε, ώστε να γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις όταν εισέρχονται τέτοια προϊόντα ζωικής προέλευσης ή γαλακτοκομικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και συχνότητα των ελέγχων προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία για τους επίσημους ελέγχους. Για τα προϊόντα κρέατος είναι το 20% απέτηση και για τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα, και το, τα πουλερικά 50% είναι το ποσοστό ελέγχων. Πρέπει να ανοίξουν δηλαδή τα φορτικά και να γίνουν έλεγχοι στα προϊόντα. Οπότε και εκεί το κόστος ε, της συμμόρφωσης της κανονιστικής θα είναι μεγάλο. Θα έχουμε επίσης καθυστερήσεις στις μεταφορές, ιδιαίτερα όταν γίνονται μεταφορές ε, ζωικών προϊόντων ή γαλακτοκομικών μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των υπόλοιπων 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα επιπλέον σημείο που ίσως δεν είχε εκτιμηθεί ιδεόντως ή ε, είναι η η αύξηση του κόστους για τις οδικές μεταφορές. Μέχρι στιγμής οι εντό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, χρησιμοποιούν μια κοινοτική άδεια. Οπότε ο, ο οδηγός μπορεί να κυκλοφορήσει ε, με την ταλίκα του χωρίς επιπλέον εμπόδια. Αν όμως ε, φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές, θα επανέλθουμε σε μια κατάσταση που ισχύει για τους Τούρκους, για παράδειγμα, οδηγούς που θέλουν να μεταφέρουν από την Τουρκία προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί οι δαλικέριδες ε, υπάγονται σε ένα σύστημα διμερών ε, ποσοστώσεων. Οπότε θα πρέπει να έχουν διαπραγματεύσεις με κάθε επιμέρους χώρα ε, για το δικαίωμά τους να εισάγουν συγκεκριμένο αριθμό φορτηγών ετησίω. Και αν ισχύσει κάτι τέτοιο και για το Ηνωμένο Βασίλειο θα αυξήσει κατά πολύ το κόστος και τα προβλήματα στις οδικές μεταφορές μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος το θέμα των Ιρλανδικών συνόρων, του Ιρλανδικού συνόρου. Ε, φυσικά η Ιρλανδία είναι η χώρα που θα επηρεαστεί περισσότερο από το Brexit. Και εδώ έχουμε δύο ε, συναφή θέματα. Το ένα αφορά το εμπόριο εντός της νήσου της Ιρλανδίας, ε, μεταξύ Βορείου Τμήματο και Ιρλανδίας, Δημοκρατία Ιρλανδίας, γιατί έχουμε πολλά ζωντανά ζώα που πάνε στη Βόρεια Ιρλανδία για να σφαγούν, ενώ εισάγονται αρνιά από τη Βόρεια Ιρλανδία. Επίσης έχουμε σημαντικές ε, μετακινήσεις νοπού γάλακτος από το βορρά προς το νότο. Εκεί οι κανονιστικέ απαιτήσει είναι μείζον ζήτημα. Τι θα, γίνει, τι θα ισχύει στις μετακινήσεις αυτών των προϊόντων. Ένα κρίσιμο θέμα και πολύ ακαθόδες. Ε, και δυσεπίλητο ε, που θα πρέπει να το συμφιλιώσουμε ως προς υποχρεώσεις και της Βρετανικής και της ε, Ευρωπαϊκής πλευράς. Σε περίπτωση που έχουμε σκληρό σύνορο με συγκεκριμένες υποδομές ηλικίες θα είναι δύσκολο. Αλλά δεν είναι μόνο το σύνορο με την Ιρλανδία, είναι γενικά το θέμα των προϊόντων που θα εξάγονται από την Ιρλανδία προς τις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες, αγορές, που ε, εξυπηρετείται κατά τον καλύτερο τρόπο από τη λεγόμενη ε, στερεά γέφυρα μέσω του, της νήσου της Βρετανίας. Καταρχάς στη, διασχίζουν δηλαδή τα προϊόντα την ε, θάλασσα της Ιρλανδίας, κατεβαίνουν στον Ντόβερ και από εκεί πάνε στη Ζεμπρούχε. Είναι το πιο οικονομικό και σύντομο μέσο, ενώ αν έπρεπε από την Νότια Ιρλανδία να περάσουν στην Γαλλία και από εκεί τη Ζεμπρούχε θα χρειάζονταν τριπλάσιο χρόνο. Άρα δεν ε, υπάρχει εναλλακτική οικονομική ως προς την οδό αυτή του εμπορίου. Ε, επίσης, και δεδομένου ότι θα περνούσαν από ένα ευρωπαϊκό μη ευρωπαϊκό κράτος, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πει ότι θα ε, προσχωρούσε στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διαμετακόμισης και άρα θα έπρεπε να έχουν τα φορτηγά το σύμβολο TIR, θα βλέπουμε πλέον ε, τέτοια φορτηγά στους ε, βρετανικούς αυτοκινητοδρόμους, αλλά πάλι δεν είναι λύση αυτή. 670 σελίδες είναι το έγγραφο το τελωνιακό το οποίο εξηγεί πώς, λειτουργεί αυτή η σύμβαση για την διαμετακόμιση, το transit και αυτό δεν αποτελεί όπως καταλαβαίνετε λύση από μόνο του, δηλαδή χρειάζονται επιπλέον διαδικασίες. Ταυτόχρονα υπάρχουν τρόποι να περιοριστούν ε, οι επιπλέον αυτές επιβαρύνσεις και εδώ σας δίνω κάποιες ιδέες, μπορεί να προκύψει δηλαδή μια τελωνιακή συμφωνία, οπωσδήποτε ευκταία αυτή καθεαυτή και βέβαια θα περιόριζε και τα θέματα της, ε, της τεκμηρίωσης, δηλαδή θα υπήρχαν τα ηλεκτρονικά έγγραφα, η προέγκριση κτλ. Αλλά αυτό δεν εξαλείφει την ανάγκη για τελωνία και ελέγχους και βέβαια και σε ε, αντίστοιχα σύνορα που έχουμε ε, με την Ελβετία, η Γερμανία με την Ελβετία ή η Σουηδία με την Νορβηγία υπάρχουν αντίστοιχοι έλεγχοι. Ε, η επανασαγωγή τώρα δασμών σε εμπορικά προϊόντα συμπεριλαμβανομένων και των γεωργικών ή, προϊόν, ή τροφίμων υπάρχει, αλλά υπάρχει και άλλη απέτηση. Οι κανόνε προελεύσεω. Μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών λοιπόν θα πρέπει να συνοδεύεται από, από κανόνε προελεύσεω. Για να κοιτάξουμε τι συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών που έχει συνάψει είτε με τον Καναδά πρόσφατα ή το Ηνωμένο Βασίλειο, μπορεί να είναι 200 σελίδε συμφωνία και μόνη αυτή καθεαυτή και 900 το κομμάτι που αφορά την ονομασία προελεύσεω. Τεράστια σημασία λοιπόν, αλλά και βαρύτητα αυτέ ε, οι συμφωνίε για το πώ ορίζεται ο τόπο προελεύσεω του, του προϊόντο το οποίο προκύπτει ε, προέρχεται από ένα κράτος. Μπορεί να υπάρχει ένα δεύτερο στάδιο τέτοιου είδους ε, κανόνων με βάση μια τακτική συνεργασία στην οποία αποσκοπούμε με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά τον Brexit. Και άλλα βήματα βέβαια ή επίπεδα ρυθμιστικής συνεργασίας με απλούστερο και πιο προφανές αυτό που είχαμε και με την ε, συμφωνία TTIP, την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών και τη δέσμευση ότι θα ε, διαβουλεύονται με αρμόδιες αρχές της άλλης χώρας αν πρόκειται να εισαχθούν νέοι κανόνες ε, που θα περιόριζαν ενδεχομένω την πρόσβαση των συντελεστών του εμπορίου, αν υπήρχαν νέοι κανόνες για το εμπόριο. Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών είναι βασικό επίπεδο συνεργασία. Μετά μπορεί να υπάρχει και αμοιβαία αναγνώριση που δεν είναι η ίδια με αυτή τη ενία αγορά. Αλλά αμοιβαία αναγνώριση που σημαίνει ότι η αρχή πιστοποίηση μιας τρίτης χώρα αναγνωρίζεται ω πιστοποιούσα το ότι το εξαγόμενο προϊόν τηρεί τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πράγμα το οποίο ιδιαίτερα σε σχέση με τα ζωικά προϊόντα το πράττουμε πολύ συχνά, δηλαδή η υπηρεσία ε, τροφίμων και κτηνιατρικών προϊόντων επισκέπτεται Φερρυπίν μια εγκατάσταση στην Βραζιλία, την πιστοποιεί και άρα αναγνωρίζει τη δική της πιστοποίηση ως αποδεκτή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι λοιπόν ζητήματα που, λύσεις που διευκολύνουν το εμπόριο, χωρίς ωστόσο να φτάνουν σε ε, ίδιες ρυθμίσεις και για τους δύο εμπορικούς εταίρους στις δύο χώρες. Επίσης υπάρχει η ισοδυναμία ρυθμιστική. Ένα επίπεδο πιο πάνω και το υψηλότερο επίπεδο, το ύψιστο επίπεδο, η εναρμόνιση που σημαίνει ότι έχουμε την ίδια νομοθεσία ακριβώς, τις ίδιες διατάξεις, όπως επίσης την ε, Γενική Συμφωνία με την Ουκρανία για τα βιομηχανικά προϊόντα. Η ισοδυναμία αναγνωρίζεται, παραμένει για τα υγειονομικά και φυτοϊγειονομικά μέσα στον ΠΟΕ και σημαίνει ότι εφόσον συμφωνήσουν οι δύο χώρες, οι δύο εταίροι, η νομοθεσία και ο τρόπος με τον οποίο εμφαρμόζεται σημαίνει ότι φτάνει στο ίδιο αποτέλεσμα ασφάλειας των τροφίμων ακόμη και αν οι προσεγγίσεις είναι κάπως διαφορετικές. Και είναι σημαντικό εδώ να, σημα... να επισημάνουμε ότι τέτοιου είδους συμφωνία ρυθμιστικής ισοδυναμίας πέραν του Ευρω... των χωρών του ΕΟΧ και της Ελβετίας που έχουν ουσιαστικά υιοθετήσει τις δικές μας ε, ρυθμίσεις, άρα πρόκειται για εναρμόνιση περισσότερο παρά ισοδυναμία, έχουμε μόνο με τη Νέα Ζηλανδία για τα ζωικά προϊόντα. Και μάλιστα ε, αναβαθμίστηκε αυτή η συμφωνία το 2015, επικαιροποιήθηκε καλύτερα με την αναγνώριση μιας σειρά από ζωικά προϊόντα και γι' αυτά λέμε ότι όντως η Νέα Ζηλανδία έχει μέτρα δύναμα με αυτά τα οποία ε, έχουμε και επιβάλλουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως και παρόλα αυτά η Νέα Ζηλανδία υφίσταται τον έλεγχο σε σημεία εισόδου και τελωνιακές άλλε επιβαρύνσει που όμω είναι χαμηλότερε, είναι πιο περιορισμένε από ότι για άλλους εταίρους. Μου επισημαίνει ο πρόεδρο ότι έχει λήξει ο χρόνος μου, επιτρέψτε μου να περάσω πολύ γρήγορα σε ένα-δύο ακόμη σημεία. Ε, το ζήτημα της ε, μετάβασης που είναι και η ουσία του προβληματισμού μας, τα τρία θέματα που μας ε, απασχολούν περισσότερο είναι η απουσία προετοιμασίας των τελωνιακών και υγειονομικών υπηρεσιών, η απουσία γνώσεως για τις χιλιάδες των επιχειρήσεων και κυρίως των μικρομεσαίων που θα εκτεθούν σε τελωνιακή διεκπαιρέωση πολύ γρήγορα και βέβαια η η μεγάλη σώρευση ε, διαδικασιών, ε, ο συνοστισμός διαδικασιών στα τελωνία που θα ξεκινήσει πάρα πολύ γρήγορα μετά το Brexit. Τι πώς θα μπορούσαν να αποφευθούν λοιπόν αυτά για μια μελλοντική ε, σχέση. Καταρχάς, θα μπορούσαν να συμφωνήσουν πριν από την 1η Μαρτίου 2019, αλλά με μια ημερομηνία λήξης ε, μιας μετάβασης ε, σε μεταγενέστερο ε, στάδιο, πράγμα το οποίο θα είναι δύσκολο και για, το, για την κυβέρνηση αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα σήμαινε ότι θα είχαμε έναν εταίρο όχι πάντα ευπρόσδεκτο και για τις ευρωεκλογέ του 2019 και για τον προσδιορισμό του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο μετά το 2020 και ούτε καθεξής. Με αποτέλεσμα όμως ουσιαστικά πως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ηνωμένο Βασίλειο από κοινού ομόφωνα θα συμφωνούσαν ε, την παράταση της ε, περίοδου των διαπραγματεύσεων. Άρα θα διατηρούνταν το, ε, το εμπόριο μόνο και μόνο επειδή το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δεύτερη επιλογή, όπω έχει πει το Ηνωμένο Βασίλειο και όπω δηλώνει ότι επιθυμεί, αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Μάρτιο του 2019, όμω βρίσκουμε έναν τρόπο για παράταση του κεκτημένου και επέκτασή του στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη μεταβατική περίοδο. Το πώς θα γίνει αυτό είναι θέμα των νομικών. Κάποιοι λένε ότι θα μπορούσε το Ηνωμένο Βασίλειο να ενσωματωθεί στον ΕΟΧ, το οποίο βρίσκω εγώ προβληματικό και το έχω αναλύσει στην μελέτη. Αλλά θα σήμαινε και περισσότερα από ότι απλώς ένταξη στον ΕΟΧ, γιατί ο ΕΟΧ δεν συνιστά τελωνιακή ένωση. Επομένω, θα έπρεπε να εξασφαλίσει τουλάχιστον μια προσωρινή τελωνιακή ένωση στο Ηνωμένο Βασίλειο και μάλιστα δεν θα καλυπτόταν καν ε, τα γεωργικά προϊόντα για ένα ελεύθερο διμερές εμπόριο. Άρα δεν είναι αυτή η λύση αποτελεσματική. Και το πραγματικό ζήτημα για μένα θα ήταν αν υπάρχει δυνατότητα σε, ένα ήδη, σε μια ήδη πολύ περίπλοκη διαδικασία διαπραγματεύσεων και για την αποχώρηση και για τις μελλοντικέ σχέσεις να την επιβαρύνουμε τη διαδικασία αυτή και με μια διαφορετικού τύπου μεταβατική περίοδο για την ε, ε, μετάβαση αυτή. Αυτά τα ζητήματα γύρω και βέβαια για τη δική σας την Επιτροπή προς διευκρίνηση παραμένουν. Το εάν θα επιτραπεί το ελεύθερο εμπόριο με το Ενωμένο Βασίλειο σε προϊόντα γεωργικά και τρόφιμα κατά τη μεταβατική περίοδο και αν συμβεί αυτό, εάν το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορέσει να παραμείνει μέλος της κοινή γεωργικής πολιτικής, εάν ενδεχομένως να παραμείνει το ελεύθερο εμπόριο με ανεξάρτητη γεωργική πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου μετά το 2019. Η οικονομική ε, διάσταση ε, βέβαια δεν μπορώ να την ε, εξαντλήσω, αλλά θα σας πω το εξής, ότι εάν προκύψει χειρότερη, το χειρότερο σενάριο, ασφαλώς θα υπάρχουν πολλά, πολλές συνέπειες, οι εξαγωγές ε, προς το Ηνωμένο Βασίλειο θα περάσουν πλέον στην ευρωπαϊκή αγορά. Ε, δύο θέματα κυρίως με απασχολούν εδώ στο τελευταίο κεφάλαιο της μελέτης. Τα μέτρα προστασίας του εισοδήματος των παραγωγών, βράχει πρόθεσμα, έχει βέβαια αρκετή εμπειρία από τα τελευταία δύο-τρία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διαχείριση κρίσεων στον τομέα τη γεωργίας, ύστερα από το εμπάργο εναντί τη Ρωσία, την κρίση στα γαλακτοκομικά. Άρα δεν ε, έχουμε τίποτε το καινούριο, ουσιαστικά επαναφέρουμε μέτρα που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί, ξέρουμε ότι είναι διαθέσιμα και μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα σενάριο ε, μετά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου. Ωστόσο, το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι δεν θα είναι προσωρινό ή κυκλικό το φαινόμενο, θα είναι μια διαρθρωτική αλλαγή αυτή της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου. Άρα θα πρέπει να βοηθήσουμε τους ε, παραγωγούς να προσαρμοστούν σε μια διαρθρωτικά διαφορετική κατάσταση τι είδου προσαρμογή των συστημάτων, τι είδου χρηματοοικονομικά μέσα, τι είδου πολιτική προαγωγή ε, θα πρέπει να προσφερθεί και τι είδου πρόσβαση σε αγορέ τρίτων ε, χωρών βεβαίω. Αυτά ευχαριστώ για την προσοχή σα. Χρειάστηκε να υπερβείτε λίγο το 20 λεπτό, εν πάση περιπτώσει. Ο κύριος Δεκάστρο, καθηγητής, ε, θέτει ερώτηση σε καθηγητή. Eh, Βεβαίω σας ευχαριστώ ιδιαίτερος και ταυτόχρονα και τους λοιπούς ε, πυρογνώμονες που μας παρουσίασαν τις τόσο ενδιαφέρουσες αυτές ε, μελέτες. Αγαπητοί συνάδελφοι, όσο προχωρούμε, όσο μελετούμε, όσο ενημερωνόμαστε για τις συνέπειες του Brexit, τόσο περισσότερο αντιλαμβανόμαστε τις τραγικές εξελίξεις που μας περιμένουν, ιδιαίτερα τους Βρετανούς βέβαια πολίτες, αλλά και πολλούς Ευρωπαίους όπως είδαμε και βέβαια τις εκμεταλλεύσεις γεωργικές και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ε, τροφίμων. Ένα γεγονός νομίζω μπορεί να περιγράψει συνθετικά την κατάσταση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αντιστοιχεί στο 7 περίπου της 100 των εξαγωγών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ η Ευρώπη εκπροσωπεί το 46% των εξαγωγών του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό είναι γεγονός, είναι δεδομένο και αναμφίβολα θα υπάρξει σοβαρή συνέπεια, σοβαρή επίπτωση, ανεξαρτήτως της όποιας πολιτικής βούλησης. Και επίσης, μια και τα ερωτήματα βεβαίως είναι επιτοπλίστων πολιτικά, ίσως δεν μπορούμε να τα διατυπώσουμε προς τους εμπειρογνωμονές μας, ε, οι τεχνοκράτες. Αλλά η συμφωνία που μπορεί να συνάψει το Ηνωμένο Βασίλειο με τρίτε χώρε είναι μια ε, πτυχή που ήδη αναφέρατε και εσείς. Δηλαδή το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να επαναδιαπραγματευτεί εξ αρχή κάθε διεθνή συμφωνία που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα σε αυτή την ε, επαναδιαπραγμάτευση θα περάσουν όλα τα θέματα. Προδιαγραφές ποιότητας, ε, προδιαγραφές ε, ευημερίας των ζώων, όλα αυτά, όλες οι συμφωνίες που έχει συνάψει η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τύχουν επαναδιαπραγμάτευσης, δεν υπάρχει εμφιβολία, δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα και βέβαια προβοκατόρικη ερώτηση προς τον φίλο Μάθιου. Μπορεί το Ηνωμένο Βασίλειο στο μέλλον να μετατραπεί σε σημείο πρόσβασης των προϊόντων που ενδεχομένως στη συνέχεια να δυσκολεύονται να μπουν στην ευρωπαϊκή αγορά. Δηλαδή αν δεν τηρούνται οι προδιαγραφές ποιότητας, οτιδήποτε απαιτούμε εμείς κατά την σύναψη συμφωνιών, διεθνών συμφωνιών με τον Καναδά ή άλλες χώρες, ε, της διεθνούς αγοράς μπορούν για το Ηνωμένο Βασίλειο να αποτελέσουν έναν επιπλέον κίνδυνο. Ευχαριστώ, Αγγουλέρα. Δεν είχα ζητήσει το λόγο. Και δεν έχουμε και πολύ χρόνο αν κάποιος τον έχει ζητήσει και θέλει να λάβει το λόγο να μην... Γιατί μας έχουν μείνει λίγα λεπτά. Εντάξει, τότε εσείς αργότερα. Ο κύριος Άγνιο. Εσείς αργότερα κύριε Κιλέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ καλή παρουσίασή σας με κάποιες πρακτικές σκέψεις. Αυτό χρειάζεται τέσσερα σημεία. Σημειώστε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει προτείνει δύο πιθανά μοντέλα, ένα απλό και μια εταιρική σχέση και φαίνεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ξέρει πώς να λειτουργήσει την εταιρική σχέση. Ε, το κάνει ήδη στην ε, νήσο του Μάν, δεν ξέρω. Ίσως πρέπει να το επισημάνω. Κάτι άλλο το οποίο δεν έχει συζητηθεί σήμερα το πρωί το Βασίλειο τώρα θα συλλέγει δασμού εισαγωγών από τρίτε χώρε. <coughs> δεν έχει συζητηθεί όμως ο οικονομικός αντίκτυπος. Βεβαίως αυτή τη στιγμή το δίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση αναφέρθηκε το κόστος εκαθάρισης αλλά τα πράγματα προχωράνε. Πριν από πέντε χρόνια όταν ε, ήθελα να οδηγήσω το αυτοκίνητό μου κατά μήκος του τάμεση, πλήρωνα σε διόδια. Τώρα το διαβάζει μια κάμερα και μου στέλνει το λογαριασμό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η τεχνολογία για να σχίσει ομαλή η ροή των εμπορευμάτων. Και τέλος μπορούμε να πούμε ότι θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος αν ξέρουμε το τι θα γίνει στο τέλος. Ε, και δεν θέλουμε να είμαστε περίεργοι. Από την άλλη ναι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ε, ένας ε, τρόπος για να παραταθεί η κατάσταση και στο μέλλον. Και ο πατέρας μου μου έλεγε «Σιουαρτ, ουδέν μονιμότερον του προσωρινού». Κύριος Άντρια. Άντρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, βέβαια, όντως, ε, η μεταβατική περίοδος που διαρκεί επαόριστον ε, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί απέναντι της. βέβαια, τα χρονοδιαγράμματα είναι πολύ σημαντικά ενώπιόν μας και για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Έχουμε πολλά χρονοδιαγράμματα μπροστά μας. Πώς μπορούμε λοιπόν να να θεσπίσουμε το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο με όλα αυτά που μας παρουσιάσατε. Γιατί σε ό,τι αφορά το ΠΔΠ και την ΚΑΠ υπάρχει το θέμα το χρονικό, το προσωρινό. Και θα εξαρτηθεί τι διάρκεια θα έχει, 5, 7 ή 10 χρόνια το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Εμείς εδώ και καιρό ζητούμε μέσω και μακροπρόθεσμες προοπτικές. Ε, και είμαστε υπέρ ε, των δεκαετών προοπτικών μάλιστα. Να έχουμε ακόμη πιο μακροπρόθεσμα ορίζοντα με διάμεση φυσικά αξιολόγηση. Τώρα, δεν μπορούμε το Brexit να το εξετάζουμε τελείως απομονωμένα. Είναι αδύνατο ε, όμως ταυτόχρονα να μπερδεύουμε και τις δύο προσεγγίσεις. Αν είχαμε μόνο βραχυπρόθεσμα προγράμματα, εντάξει. Αλλά πώς είναι δυνατόν να εμπλέξουμε την Ευρώπη σε μία ε, επταετή, δεκαετή προοπτική χωρίς να έχουμε προηγουμένως διευθετήσει το ζήτημα του Brexit. Αυτό δεν το κατάλαβα από τη μελέτη σας. Και πάλι θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μαθιού για την εξαιρετική ε, παρουσίαση και, και μία ώρα να μιλούσατε θα σας άκουγα. Λοιπόν, για το πού θα πάει το τυρί μας εάν δεν μπορούμε να το στείλουμε στη Βρετανία. Επειδή είμαι παθιασμένος με το τσένταρ και όταν είχε έρθει η οικογένειά μου τρέχαμε σε όλες τις Βρυξέλλες για να το βρούμε και διαπιστώσαμε ότι είναι ε, δύσκολο και υπάρχει λόγος. Δεν τρώνε πολύ τσένταρ εδώ, δεν τρώνε τσένταρ στη Γαλλία και πού θα το στείλουμε θα αρχίσουμε την παραγωγή μπρι και το άλλο. Και δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας. Ε, ίσως ε, δεν μπορείτε να απαντήσετε γιατί είναι και πολιτικό το ζήτημα. Βασιζόμαστε, όπως ε, ακούστηκε, ε, στην αλληλεγγύη και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους μη και Ιρλανδούς που ήρθαν σήμερα, αλλά είναι σαφές ότι εάν δεν είμαστε εμείς, δεν αφορά το ζήτημα τους άλλους τόσο πολύ. Ε, χρειαζόμαστε λοιπόν αλληλεγγύη. Πού είναι η αλληλεγγύη των άλλων χωρών και είναι εκπληκτικό ότι στο μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας, στην πιο σημαντική συνεδρίαση που είχαμε στην Επιτροπή μας για τον Brexit, να υπάρχει κανείς εδώ από την Ολλανδία. Ε, τι, τι βοήθεια θα λάβουμε αν δεν έχουν έρθει σήμερα να ακούσουν καν τα ζητήματα για να τα μεταφέρουν στην κυβέρνησή τους και να τους πούν ότι η Ιρλανδία θα έχει σοβαρό πρόβλημα. Δεν μπορούν να το κάνουν γιατί δεν είναι εδώ που είναι η αλληλεγγύη και ευχαριστώ τους παρόντες που μπορεί να μην επηρεάζονται τόσο, αλλά έχουμε έρθει να μιλήσουμε. Ορίστε, με ποιον θα μιλήσουμε. Και πληρώνονται βεβαίως αδρά. Κύριε Μαγκίνες, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία ερώτηση. Αναφέρατε τις διαρθρωτικές αλλαγές. Ε, πείτε μου, ποιες θεωρείτε ότι θα είναι οι διαρθρωτικές αλλαγές λόγω Brexit στην ε, Ευρωπαϊκή Γεωργία. Κυρία Κάντενμπαχ. Να θερμά ευχαριστώ. Θα συμφωνήσω με τα όσοι είπε ο και ίσως να μην σας ε, άκουσα και τα προσεκτικά, αλλά τέτοιου είδου μελέτες παρουσιάζονται και στην Επιτροπή των Προπολογισμών ή υπάρχει κάποια πιθανότητα, διότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που συζητούμε εδώ πέρα, είναι πολύ καλό το υλικό και θα ήταν οπωσδήποτε πολύ σημαντικό και οι συναφή της Επιτροπή των Προϋπολογισμών να έχουν την τύχη να ε, ασχοληθούν με τα ίδια αποτελέσματα και πορίσματα των μελετών σας. Ναι. Ε, βέβαια, ο πρόεδρος της ε, Επιτροπής Προπολογισμού είναι αναπληρωτής στη δική μας Επιτροπή και ε, παρακολουθεί τα θέματα, αλλά πολύ σωστά το επισημάνατε. Κύριε καθηγητά, έχετε έξι λεπτά ε, και με την επίκαια των διερμηνέων μπορείτε να λάβετε ακόμη πέντε, πέντε επιπλέον. Παρακαλώ. I think I can be uh, quicker than I was. Πιο σύντομος από ότι στην πρώτη μου παρέμβαση. Ένα, δύο, τρία θέματα έχω. Ο κύριος Δεκάστρο ρώτησε αν μπορεί να αποτελέσει μια πίσω πόρτα σε σχέση με μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου του ΕΒ. Πολλά εξαρτώνται από τους λοιπούς συντελεστές. Το πλαίσιο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί αυτό, εάν επί παραδείγματι θα μείνει μέσα το Ηνωμένο Βασίλειο στην Τελωνιακή Ένωση κατά τη μεταβατική περίοδο, αν ε, υπάρξει συμφωνία για εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου, όλα αυτά ε, προφανώς δεν μας ανησυχούν. Εάν όμως συμβούν στα τρόφιμα, κάτι που έχει συμβεί στην Ευρώπη είναι ότι εφαρμόζονται πολύ αυστηρά συστήματα ανιχνευσιμότητας. Και ξέρουμε ότι οι επιθεωρητές τροφίμων δεν κοιτούν μόνο ποια παρτίδα έχει περάσει τα σύνορα, αλλά κοιτούν τη διαδικασία και στην επεξεργασία και στο, ε, στη διάθεση στο ελληνικό εμπόριο. Κοτόπουλο, παραδείγματι. Κρέας πληρικών. Χωρίς φυσικά σύνορα στον νησί της Ιρλανδίας και με συμφωνία ελεύθερων ε, ε, συναλλαγών με το Ηνωμένο Βασίλειο, αμερικανικό κοτόπουλο θα μπορούσε να απολύεται όχι μόνο στην Ιρλανδία, βρετανικό μάλλον εννοεί ο μιλητή, όχι μόνο στην Ιρλανδία αλλά και στην, στο υπόλοιπο, στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αυτό πάλι θα ξεκριθεί από την, από την ανιχνευσιμότητα που θα έχουμε για ε, τον κύριο Άγνου. Βεβαίω, ε, λαμβάνω υπόψη τα σχόλιά του. Η εξαιρετική μελέτη που παρουσιάστηκε ω προ τι δημοσιονομικέ συνέπειε του Brexit λαμβάνει υπόψη και τι συνέπειε ω προ τα τελωνιακά έσοδα στα οποία αναφερθήκατε κι εσείς, δηλαδή θα υπάρχει αυτό το εισόδημα από την ε, ίσπραξη δασμών του Ηνωμένου Βασιλείου από τρίτες χώρες που δεν θα διαβιβάζεται πλέον στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Άρα θα υπάρχει σχετικά αύξηση των πόρων για το Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης, ε, στο συσχετισμό μεταξύ αυτής της μεταβατικής περίοδου και των διαπραγματεύσεων για την ΚΑΠ και το πολιτεύσιμο οικονομικό πλαίσιο, είδαμε ήδη ότι έχει μετακυλιστεί ε, το περιθώριο για το πουδουπού από φέτος μάλλον Περιμένουμε τώρα την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Μάιο του 2018. Θα δούμε αν υπάρξει σαφήνεια ως προς το οικονομικό σκέλος, ως προς το δημοσιονομικό σκέλος, ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν αυτές οι συνομιλίες. Αλλά προφανώς πολλές θα είναι οι χώρες οι οποίες δεν θα είναι διατεθειμένες να μπουν στη συζήτηση αυτή, εάν ακόμα παραμένει ασαφής η κατάσταση σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Συμφωνώ λοιπόν ότι είναι ασαφέστατη η κατάσταση. Κύριος Φλάναγκαν, για το Τσένταρ συγκεκριμένα. Βεβαίω μπορεί να αποτελέσει σοβαρό πρόβλημα για τους ε, παραγωγούς ε, που ασχολούνται με την κατεργασία γαλακτοκομικών προϊόντων, γιατί δεν υπάρχει κατανάλωση τόση στην υπόλοιπη Ήπειρο την Ευρωπαϊκή Ήπειρο δηλαδή του Τσένταρ, αλλά βέβαια μπορεί το Ηνωμένο Βασίλειο να βρει λύσεις με τον ΠΟΕ ώστε να μειώσει ή να βρει κοινού δασμολογικούς ε, ε, κοινέ δασμολογικέ λύσει, ε, κοινά δασμολογικά τιμολόγια ω προ τι πωλήσει προ τρίτε χώρε. Και έτσι θα πωλείται με του ίδιου δασμού το προϊόν αυτό προ τρίτε χώρε και έτσι οι Ιρλανδικές εξαγωγές προς τη ε, Βρετανία ή οι Βρετανικές εξαγωγές κρέατος προς την υπόλοιπη Ευρώπη μπορούν να καλύπτονται από τους ίδιους το ίδιο δασμολογικό τιμολόγιο. Υπάρχει βέβαια και το χειρότερο σενάριο, έτσι, και ενώ μπορούμε να έχουμε μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, μπορούμε πάλι να κάνουμε εξαγωγές από την Ιρλανδία στην ε, ε, Βρετανία του Τσένταρ χωρίς δασμούς, αλλά αν βρεθεί η καλύτερη λύση, ενώ αν υπάρχουν δασμοί, με βάση και τα χρονοδιαγράμματα του ΠΟΕ θα είναι δύσκολο, δύσκολη η επίλυση του θέματος, θα πρέπει να διαφυλαχθεί το δασμολόγιο. Για τις διαρθρωτικές αλλαγές και την κυρία Κάτνμπαχ βεβαίως υπάρχουν δύο στοιχεία, οι εξαγωγές από την Ιρλανδία με, τα πρόσθετα, με τους πρόσθετους φραγμούς της εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο σημαίνουν ότι μπορούν να βρουν λύσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πρέπει να αναζητήσουν και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, δεν ξέρω τι έχει υπόψη η Ιρλανδική κυβέρνηση. Έχει προβλέψει πάντως το προσεχή προϋπολογισμό περισσότερη χρηματοδότηση στην προβολή προϊόντων, στο μάρκετινγκ δηλαδή προϊόντων για τον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά βέβαια ξέρουμε ότι θα έχει και τα σοβαρότερα πλήγματα, η Ιρλανδική οικονομία σε αυτό θα χρειαστεί μεγαλύτερη προσαρμογή και βέβαια υποστήριξη από τα συστήματα. Πρόεδρος. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά. Καταφέραμε να ολοκληρώσουμε και στην ώρα μας. Ευχαριστώ θερμότατα τους καλεσμένους μας, τους εμπειρογνώμονες για τις πολύ ενδιαφέρουσες μελέτες τους θα έχουμε το χρόνο με την ησυχία μας να διαβάσουμε και αναλυτικά τις εκθέσεις. Και πιστεύω ότι σήμερα είναι η αρχή μιας σειράς παρόμοιων συζητήσεων που θα γίνουν και στο μέλλον, γιατί υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες και σαφή σημεία. Και νομίζω θα πρέπει να βρούμε άλλη μορφή συνεργασίας μία άλλη μορφή συνεργασία που θα είναι αμοιβαίω επωφελή. Νομίζω ότι όλοι θα χρειαστεί στις διαπραγματεύσεις να κάνουμε παραχωρήσεις, χάρη συμβαστικής λύσης. Θα πρέπει να διατυπώσουμε τις προσδοκίες μας, να εκθέσουμε τις απόψεις μας, να αξιοποιήσουμε τα κονδύλια μας. Δεν θέλουμε να βρεθούν κερδισμένοι και χαμένοι. Θέλουμε μια συμφωνία που θα είναι επωφελής και για τις δύο πλευρές. Κάτι που θα είναι μάλλον δύσκολο, μια τέτοια συμφωνία θα είναι αρκετά δυσέβρετη, αλλά αυτό είναι ο στόχος μας. Σας ευχαριστώ και πάλι θερμά για τη συμμετοχή. Ραντεβού στις 13 Νοεμβρίου στο Στρασβούργο, 7 με 10 και μισή. Μετά θα έχουμε συνεδρίες 22 Νοεμβρίου πρωί και απόγευμα, 23 Νοεμβρίου ε, το πρωί και 29 Νοεμβρίου το βράδυ, 7 με 9.30. Παρουσία του Επιτρόπου Χόγκαν, που θα μας κάνει την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα μας την παρουσιάσει. Ε, έχουμε συνεδριάσεις και το Δεκέμβριο. Έχουμε αρκετέ τον Εύρο, αλλά έχουμε και το Δεκέμβριο. Ευχαριστώ θερμά, ιδιαίτερα όσου άντεξαν μέχρι το τέλος. Ευχαριστώ τους ειδικού μας, τους εμπειρογνώμονές μας, τους συναδέλφους. Σας ευχαριστώ πάντως που πραγματικά εμπλουτίσατε τις συζητήσεις μας και σας εύχομαι καλό απόγευμα σε όλους και στους διερμηνείς. Κυρίσω το πέρας συνεδρίασης.